Oh, if you take your Παρακαλώ καθίστε, μπορούμε να ξεκινήσουμε. thank you Ευχαριστώ πολύ. Ε, ξέρω ότι δεν είναι και τόσο βολικό να βρισκόμαστε σε αυτή την αίθουσα, αλλά υπήρχε μια ομάδα μαθητών που τους δώσανε την άδεια να έρθουν στο ημικύκλιο και γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ. Όπως θα παρατηρήσετε, δεν μπορούμε να πιούμε κάτι εδώ μέσα. Είδα κάποιος που μπορεί καμιά φορά να βάζουν μέσα κρυφά, αλλά έξω υπάρχουν καφέδες και οι κλητήρε δεν θα σας αφήσουν να τους βάλετε μέσα. Κάποια στιγμή θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα, οπότε όσοι θα είναι παρόντες όλη την ώρα της συνεδρίασης θα μπορέσουν να πιουν λίγο καφέ. Ωραία. Λοιπόν, τώρα φτάσαμε στο σημείο 6 και 7 τη ημερήσιας διάταξή μας, ε, που είναι η εξέταση των ε, τροπολογιών για το ΜΥΦΙΤ και το Νιφέρ και θα δώσω τον λόγο στον Μάρκους Φέμπερ, τον εισηγητή. Μάρκους. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να πω στους ε, μαθητές ε, ότι είναι καλό που τους έχουμε εδώ. Καταρχάς να πω ότι έχω ε, στο σωστό χρόνο και με επαρκή χρόνο τη δυνατότητα να μιλήσω για αυτό το πολύ δύσκολο θέμα της ρύθμισης της αγοράς. Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία αναλάβαμε σε αυτή την ε, νομοθετική περίοδο, μια γενική, δηλαδή ρύθμιση της αγαράς. Ε, πρέπει λοιπόν να σας θυμίσω ότι στο Πίτσμπουργκ ε, συμφωνήθηκε στο G20 τα κράτη να έχουν γενικές ρυθμίσεις ώστε να μην υπάρχει καμία αρρύθμιστη αγορά ή ε, χρηματοπιστωτικά προϊόντα ε, αρρύθμιστα. Αυτό λοιπόν ε, ξεκίνησε μια νέα ευκαιρία στο Pittsburgh την οποία τώρα εμείς πρέπει να κλείσουμε με πολύ προσοχή παρακολουθούμε αυτά που γίνονται στο Μεξικό ε, και είναι σωστό αυτό γιατί ως Ευρωπαϊκή Ένωση εμείς συμβάλλουμε ε, πολύ στη σταθεροποίηση της χρηματοπιστωτικής αγοράς. Θα πρέπει όμως και να προσέχουμε όταν ε, έχουμε πολύ αυστηρούς κανόνες να προσπαθούμε να μην εξασθενήσουμε τις δικές μας αγορές ε, και οι άλλες ε, που δεν είναι ρυθμισμένες να ενδυναμώνονται. Να μιλήσω τώρα για κάποια συγκεκριμένα σημεία. Πραγματικά με εξέπληξε με ποια φέλια από τη μία πλευρά και με ε, ποια προσπάθεια να βελτιωθεί ο κόσμος των χρηματοπιστωτικών προσπάθησαν οι διάφορες ομάδες ενδιαφερόντων να επηρεάσουν. Και δεν εννοώ το λόμπι των τραπεζών που υπάρχει. Αυτοί θέλουν να βελτιωθεί ε, ο κόσμος τους και καταθέτουν ε, ζητήματα και ε, μπορεί να κάνουν και δραστηριότητες που δεν είναι πλέον αποδεκτές και θα επανέλθω σε αυτό το θέμα γιατί σε κάθε συζήτηση το λέω και νομίζω ότι και οι συνάδελφοι ε, το έχουν παρατηρήσει. Ε, υπάρχει στο Στρασβούργο, ας πούμε, περίπτωση να μου τεθεί ερώτηση η οποία δεν έχει καν σχέση με την πραγματικότητα. Όταν με κατακλείζουν με email ε, που είναι αντικειμενικά λάθος ως αντιλήψεις, πραγματικά ειλικρινά, δεν ξέρω αν μπορώ να είμαι πιο συμβιβαστικός ε, από ό,τι ήμουνα στις διαπραγματεύσεις. Γιατί δεν υπάρχουν άλλες ε, ε, δυνατότητες από αυτές που έχω ήδη δείξει. Αυτά για τα γενικά στοιχεία. Πάμε τώρα στα θέματα. Σημείο 1. Ε, εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής. Ε, στο G20 ε, μας θεσπίστηκε η υποχρέωση να μην υπάρχουν μη ρυθμισμένες αγορές και προϊόντα. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, όταν πάμε στο χρηματιστήριο στις Βρυξέλλες, υπάρχουν τουλάχιστον για μένα τουλάχιστον δύο ε, χαρτιά τα οποία σήμερα δεν είναι ρυθμισμένα. Το ένα είναι οι μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, ε, τράπεζες, συγγνώμη, οι οποίες ε, στο μέλλον θα πρέπει να μπίπτουν στο ΜΥΦΙΤ. Και πραγματικά δεν ξέρω ή κανείς να μου πει γιατί γίνεται αυτό. Ξεκάθαρα φαίνεται ότι ε, δεν μπορεί ε, το, ο Ευρωπαίος Νομοθέτης ε, να αφήνει μια τρύπα η οποία ε, τελικά ναι μεν στην αρχή θα λένε ότι δεν δημιουργεί προβλήματα αλλά μετά θα βγαίνει ένα θυγατρικό εμπόρευμα ας πούμε το οποίο θα δημιουργεί πρόβλημα. Έτσι λοιπόν στην πραγματική οικονομία ε, θα πρέπει να υπάρχουν ε, χαρτιά τα οποία θα ε, είναι ρυθμισμένα και δεν θα υπάρχουν μεγάλες εξαιρέσεις. Εξαιρέσεις και σε αυτόν τον τομέα. Όμως θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό που πραγματικά θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις. Ε, και όποιος εδώ ε, βλέπει ότι υπάρχει ε, μια μεγάλη εξαίρεση, όποιος δημιουργεί μια μεγάλη εξαίρεση, στην ουσία δημιουργεί μια μεγάλη τρύπα, μια μεγάλη πύλη, η οποία θα αποτελέσει κερκόπορτα για την ρύθμιση της αγοράς. Γι' αυτό θα πρέπει να προσπαθήσουμε μαζί με τους ε, συναδέλφους να έχουμε τόσο μικρές τρυπούλες ε, όσο δυνατόν γίνεται. Ε, να επικεντρωθούμε σε αυτό που είναι πολύ σημαντικό. Δεύτερο θέμα, διάρθρωση της αγοράς. Νομίζω ότι αυτό είναι η μητέρα όλων των ζητημάτων. Γιατί έχει να κάνει με την ρύθμιση της κατάχρησης της αγοράς. Και το έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα. Έχουμε εδώ μια πρόταση της Κομισιόν να υπάρχει άλλο ένα χαρτί που ονομάζεται Οργανωμένοι Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης. Ε, ε, μέσα από αυτό θα μπορέσουμε να ε, ενισχύσουμε τις δομές έτσι ώστε να βελτιωθεί η ρύθμιση της αγοράς και υπάρχουν και άλλες τροπολογίες που δεν θέλουν καθόλου να επιτραπεί. Σας λέω ξεκάθαρα ότι δεν μπορούμε να έχουμε συμβιβασμούς σε κατεύθυνση είτε UTF είτε όχι UTF είτε το ακολουθούμε είτε όχι. Έκανα κάποιες συζητήσεις με τους σκιώδεις και δεν μπορέσαμε να συμφωνήσουμε. Εγώ προσωπικά από το σχέδιο ε, κατά, διαβάζοντας το σχέδιο της πρόταση, θεωρώ ότι αυτά τα, αυτοί οι οργανωμένοι μηχανισμοί διαπραγμάτευσης είναι κάτι σωστό, είναι μια, ε, ένα συμβιβασμός μεταξύ των διαφόρων θέσεων. Ελπίζω να βρούμε μια λύση, γιατί αυτό το θέμα ε, δεν έχει ξεκαθαρίσει μεταξύ των διαφόρων ομάδων και θα είναι δύσκολο όλο το πακέτο να το αντιμετωπίσουμε χωρίς αυτό. Ένα άλλο θέμα ε, το οποίο μας ανησυχεί, το οποίο αμένα όχι τόσο θα έλεγα, είναι η προστασία των επενδυτών. Ο δρόμος που πρότεινε η Κομισιόν είναι ε, πολύ πιο απλός. Η Κομισιόν λέει ότι υπάρχει ανεξάρτητη παροχή συμβουλών που ακολουθεί κάποια συγκεκριμένα κριτήρια ε, και υπάρχουν και οι υπόλοιπε συμβουλές που δεν τις ρυθμίζουμε. δεν πρέπει να πάμε έτσι θα πρέπει να φροντίζουμε τους πελάτες και τις ανάγκες τους για συγκεκριμένα ε, προϊόντα και αυτό ε, ε, δεν έχει να κάνει με τους επαγγελματίες, ας πούμε, επενδυτές, έχει να κάνει με τους μικρούς, τους μη επαγγελματίες. Το λέω ήδη ότι δεν μπορεί ο Ευρωπαίος νομοθέτης να έχει ως έργο να αλλάζει δομές ο οποίος δεν έχει επαληθεύσει ότι είναι λάθος. Ε, υπάρχει λοιπόν ε, πολλές φορές αυτή η προσέγγιση και τελικά δεν ρυθμίζεται το πρόβλημα. Και αυτό μου λέει η Κομισιόν ότι θέλει να αλλάξει κάποιο πρόβλημα ε, και δεν προτείνει κάποιες ε, γενικές απογορεύσεις διατάξεων. και προμηθειών. Ε, πρέπει να δούμε τι θα γίνει ε, ε, με το θέμα των προμηθειών. Έχουμε κράτη-μέλη που δεν το κάνουν αυτό. Έχουμε κράτη-μέλη όπου έχουμε την κουλτούρα του ανεξάρτητου συμβούλου και άλλα στα οποία δεν υπάρχουν. Υπάρχει υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη τα οποία ε, μας λένε ότι εδώ ε, η λέξη κλειδί είναι μόνο η επικορικότητα. Δηλαδή να αφήσουμε τα, την αγορά να ρυθμιστεί μόνη της. Και αν θέλουμε τώρα να φέρουμε και διαφάνεια στην αγορά, αυτό είναι ξεκάθαρο. Τότε θα πρέπει να υπάρχουν προβλέψεις. Υπάρχουν πολλές τροπολογίες που πηγαίνουν ε, προς αυτή την κατεύθυνση να προστατεύσουμε τους καταναλωτές και ευχαριστώ τους συναδέλφους ε, που μιλήσαμε για αυτό το θέμα πάρα πολύ και έχουν καταφέρει να καταθέσουν μια πολύ καλή λύση η οποία από τη μία πλευρά ε, λαμβάνει υπόψη ότι η Ευρώπη έχει τον πλούτο της ποικιλία και από την άλλη κοιτά ότι η πελάτες και συγκεκριμένα οι μικροί επενδυτές ε, χρειάζονται κάποια προστασία. Το δεύτερο είναι το θέμα πώς μπορούμε ε, να έχουν πρόσβαση σε ε, αυτή την προστασία. Είναι το θέμα της καταγραφής των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. Λέγεται ότι θα πρέπει να υπάρχει αυτή η υποχρέωση σε όλη την Ευρώπη. Όμως τους μικρούς επενδυτές Όταν παίρνουν τηλέφωνο στην τράπεζά τους και ε, ε, λένε ότι μου περισσεύουν κάποια ε, λεφτά γιατί πήρα ένα μπόνους ή μου εξοικονόμησα κάποια χρήματα και θέλω να τα επενδύσω και αυτά καταγράφονται όλα στο τηλέφωνο, εγώ πραγματικά θεωρώ ότι τα κράτη-μέλη που το έχουν αυτό ήδη ε, ωραία, να το κρατήσουν, αλλά αυτά ε, που δεν το έχουν θα πρέπει να το κάνουν μόνο για τους επαγγελματίες. Για τους υπόλοιπου θα πρέπει να είναι επιλογή. Αυτό θεωρώ ότι είναι ο σωστό δρόμο. Άλλο θέμα έχει να κάνει ε, με το τη γενικά και με... Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι οι συναλλαγές υψηλής συχνότητας. Να πω ότι η εισαγωγή του κομπιούτερ στο πακέτο ήταν λάθος και έπρεπε να ανατραπεί. Επίσης, στο πακέτο χωρίς κομπιούτερ υπάρχουν δυνατότητες ε, κατάχρησης αγοράς. Ε, όμως υπάρχουν ε, νέες προκλήσεις με την εισαγωγή της τεχνολογίας συγκεκριμένα. Μπορεί κανείς πολύ γρήγορα μέσα από αλγορίθμους, από software να αναλύσει τι ακριβώς συμβαίνει και ε, όταν ε, ε εγώ δεν ενδιαφέρομαι για ένα προϊόν μπορεί τελικά να μην έχει μεγάλη ε, σημασία. Από την άλλη όμως επηρεάζει και την ρευστότητα στις αγορές. Να το πω ξεκάθαρα ότι αυτά τα χρηματιστήρια που ε, προσανατολίζονται στο να βγάζει κανείς γρήγορα χρήματα θα πρέπει να τους ζητηθούν να ε, κοιτάξουν τη ζήτηση, να φτιάξουν μια συγκεκριμένη ε, προσφορά τιμής και μετά να υπάρχει ένα όργανο ε, διαχείρισης το οποίο θα έχει κάποια λογική. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποια είναι η, τα καθήκοντα αυτών των πλατφορμών ε, διαπραγμάτευσης. Ε, υπάρχει και το θέμα της ε, διαπραγμάτευσης ε, των αλγορίθμων. πρέπει να βάλουμε πιο αυστηρούς κανόνες. Δεν λέμε να τα απαγορεύσουμε, αλλά να είναι πιο αυστηροί οι κανόνες. Τώρα, για τις ε, ε, διαπραγματεύσεις υψηλής συχνότητας. Είμαστε στα 5 εκατοστά του χιλιοστού. Στα αυτό τι σημαίνει, ότι κάτι ε, δίνεται και αμέσως αποσύρεται. Από αυτό ε, κανείς υποθέτει ότι υπάρχουν εντολές οι οποίες κατατίθενται ε, μόνο και μόνο για να δώσουν κάποια κατεύθυνση και να επηρεάσουν την τιμή, δηλαδή εντολές πώληση ή αγοράς. Και όταν συζητάμε για αυτά τα θέματα με τους ειδικού ε, και λέμε ότι θέλουμε να το λύσουμε μέσα από το MIFID, μας λένε ότι είναι σωστό. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει οι εντολές να παραμένουν λίγο περισσότερο ίσως. Αυτό είναι θέμα νούμερο ένα. Το θέμα νούμερο δύο. Όταν κανείς ε, η θελημαία ε, μπαίνει στην αγορά μαζικά με εντολές, τις οποίες μετά αποστήρει... Ε, χρησιμοποιεί την υποδομή ε, η οποία τελικά δεν δημιουργεί οικονομικά προστιθέμενη αξία και δεν πληρώνει και αντίστοιχα ε, τέλη. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια γενική αρχή η οποία θα λέει ότι όποιος χρησιμοποιεί πάρα πολύ την υποδομή θα, έχει και, θα πρέπει να έχει και ένα κόστος μέσα από τέλη που θα πρέπει να πληρώνει. Το επόμενο θέμα είναι θα πρέπει όντως κάθε χρηματοπιστωτικό προϊόν να δημιουργεί κάποια τιμή όταν είναι τόσο μικρή η αξία του. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε εάν ε, αυτά τα μικρά προϊόντα ε, μπορούν να επηρεάζουν τις τιμές ή όχι. Και σε αυτό το θέμα ε, υπάρχουν διάφορες τροπολογίες και ευχαριστώ τους συναδέλφους ε, που πάνε λίγο πολύ στην ίδια κατεύθυνση. Χαίρομαι ότι όταν μιλάμε για συναλλαγές υψηλής συχνότητας είναι καλό να υπάρχουν κανόνες παιχνιδιού οι οποίοι θα βοηθούν την αγορά ε, και θα μειώνουν τις δυνατότητες κατάχρησης της αγοράς. Άλλο θέμα τώρα είναι η ρύθμιση των τρίτων χωρών. Στο μεταξύ, σε αυτή την νομοθετική περίοδο έχουμε ε, ψηφίσει διάφορες, ε, διάφορες ρυθμίσεις για τα τρίτες χώρες, ε, Εναλλακτικέ ε, μορφές διαχείρισης των επενδύσεων. Ε, υπάρχει... Υπάρχουν διάφορες ρυθμίσεις, λοιπόν. Θεωρώ πρέπει να ξέρουμε ε, τι έχει να κάνει με το MIFID και τι όχι. Με το MIFID δεν μπορούμε να εμποδίσουμε έναν πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επενδύσει τα χρήματά του στο Hong Kong. Δεν μπορούμε επίση να απαιτήσουμε ε, να έχουν κανόνες μήφετ τα χρηματιστήρια στο Χονγκ Κονγκ. Είναι ε, στο πεδίο τη ρύθμιση των τρίτων χωρών. Επίση, δεν μπορούμε να, να εμποδίσουμε κάποιον από το Χονγκ Κονγκ να επενδύσει χρήματα στο Λονδίνο ε, και στο Παρίσι. Και τότε θα εμπίπτει στου κανόνες μήφετ. δεν νομίζω ότι μπορούμε μέσα από τη ρύθμιση των ε, τρίτων χωρών να αγγίξουμε τέτοια θέματα. Μόνο το ποιο έχει πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές. Υπάρχει η αρχή της αντιστοιχίας, ε, ε, equivalence principle και η αρχή της αμοιβαιότητας αμοιβαία, δηλαδή να ζητάμε να ισχύουν πράγματα, αλλά έτσι βάζουμε τα χέρια μας και βγάζουμε τα μάτια μας. Αν ε, θέλουμε να έχουμε επενδυτές από τρίτες χώρες, πραγματικά αυτή η αρχή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Θα πρέπει να αφήσουμε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, που είναι ο υπεύθυνο να ασχοληθεί με αυτά τα θέματα. Ένα άλλο θέμα ε, που ε, συζητείται πολύ έτσι ιδεολογικά είναι ε, το θέμα των ορίων θέσεων. Δεν μπορούμε να πούμε να βάλουμε ένα πολύ αυστηρό τέτοιο ε, σύστημα και εμείς είμαστε καθαροί Ευρωπαίοι, ε, νύπτουμε τα σχήρας μας, έχουμε λίστα προβλήματα και δεν έχουμε καμία κερδοσκοπία. Ε, μπορεί να γίνουν περίεργα πράγματα όταν τελικά υπάρξει κερδοσκοπία, να υπάρξει αλλά όχι με τους δικούς μου κανόνες παιχνιδιού. Και εάν μέσα από πιο αυστηρούς κανόνε τελικά καταλήξουμε ώστε να υπάρχει αυτή η κερδοσκοπία, τότε δεν έχουμε πετύχει το σκοπό μα. Να πω ξεκάθαρα ότι Ε, πραγματικά ε, άκουσα πολλές προτάσεις. Στις δικές μου τροπολογίες έχω διαχωρισμό ανάμεσα στα, ε, σε αυτούς που έχουν φυσικό ενδιαφέρον για κάποιο προϊόν και σε αυτούς που δεν έχουν. Αυτοί που δεν έχουν, ε, τότε τους υποβάλλω στο καθεστώς αυτό των ορίων θέσεων πρακτικά αυτό ε, θα μας βοηθήσει να λειτουργήσει η αγορά. Αλλά να πω, όποιος δεν έχει φυσικό ενδιαφέρον, τότε αυτός θα πρέπει ε, να υποβάλλεται σε όρια γιατί ουσιαστικά ασκεί κερδοσκοπία. Αυτοί που έχουν ενδιαφέρον, από την άλλη είπα, οι οποίοι ε, ως τώρα δεν υπόκεινται σε κανένα καθεστώς, για αυτούς ε, θα ήθελα έναν έλεγχο θέσεων, ε, δηλαδή κάνω τα πράγματα πιο αυστηρά. Να πω ξεκάθαρα λοιπόν ότι το αντίθετο είναι το σωστό. Εγώ διαφοροποιώ αυτούς που έχουν ενδιαφέρον από αυτούς που δεν έχουν και σε αυτούς που έχουν ενδιαφέρον ε, βάζω ακόμα ένα άλλο εργαλείο ε, διαχείρισης. Γι' αυτό είμαι κατά όλων των τροπολογιών ε, που ε, είναι υπέρ των over-the-counter ε, συναλλαγών, γιατί μετά έρχονται τα άλλα προϊόντα τα οποία είναι πολύ δύσκολο να ρυθμιστούν. έτσι χρηματιστηριακά προϊόντα τα οποία ε, αυξάνουν το ρίσκο και δεν, τον, ε, δεν το μειώνουν. Και δεύτερον, νομίζω ότι ο Ευρωπαίος νομοθέτης δεν μπορεί να ρυθμίσει αυτές τις αγορές εκτός της Ευρώπης, στο Σικάγο ας πούμε. Ε, μπορεί να υπάρχει ε, αντίκτυπος αν εμείς δεν έχουμε σωστούς κανόνες. Έτσι λοιπόν για μας ε, καλό θα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε κανόνες ε, που ε, θα πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση και να μην τους υποστηρίζουμε με λάθος επιχειρήματα. Υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία θα ήθελα να θίξω πολύ σύντομα. Είναι η ολοκλήρωση των δεδομένων όταν ε, ε, υπάρχουν προϊόντα ε, μη μετοχικά, θα πρέπει να πάμε πολύ γρήγορα. Συγγνώμη, λέει, η πρόεδρος διακόπτη. Η πρόεδρος διακόπτη. Αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου, είμαστε εδώ γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Σχεδόν ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι στον κόσμο υποσυτίζονται When, if you shut up, please, and would listen. Για σταματήστε για να μπορέσουμε να ακούσουμε. Okay, right. Um, I will give the floor. Ωραία. εξαιρετικός τρόπος για να προκαλέσει κανείς ε, τη δημόσια κατανόηση. Πραγματικά δεν ξέρω περί τίνος πρόκειται. Εκπρόσωποι της βιομηχανίας, ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Ο Μάρκος. Ευχαριστώ. Α, θέλετε να πάρετε το λόγο. Θέλω να συνεχίσω, λέει ο μιλητής. Κοιτάξτε, διαδικαστικό, κυρία Πρόεδρε. Δεν ξέρω, είναι σκόπιμο να εμφανίσουμε αυτή την εικόνα εδώ, σε αυτή την αίθουσα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε για ποιο λόγο βρισκόμαστε σε αυτή την αίθουσα. Υπάρχουν πάρα πολλές ε, διαθέσιμες χώρες, ε, αίθουσες. Εξήγησα την ε, προηγούμενη φορά σας είπα ότι βρισκόμαστε εδώ γιατί η αίθουσα που συνήθως χρησιμοποιούμε χρησιμοποιείται από μία ομάδα μαθητών. Γι' αυτό το λόγο μα χρειάστηκε να συνεδριάσουμε εδώ. Ο Μάρκο κάνει μια θαυμάσια παρουσίαση των τροπολογιών και πραγματικά θα ήθελα να του δώσουμε και πάλι το λόγο. Ευχαριστώ. Ωραία, συνεχίσω λοιπόν, αφού με διέκοψαν. Υπάρχουν τροπολογίες οι οποίες αναφέρονται στην απαγόρευση των υπερβολικών κερδοσκοπιών. Βεβαίως μπορούμε να δεχτούμε αυτές τις τροπολογίες, αλλά αυτό δεν είναι ιδιαίτερα θετικό. Θα μπορούσαμε να αποφασίσουμε για ένα σύστημα το οποίο θα θέτει ορισμένα όρια. Για παράδειγμα, στον ε, τομέα των ε, ειδών διατροφής στο Παρίσι, για, στον τομέα των, ε, της ε, βιομηχανίας μετάλλου στο Λονδίνο. Οι αναπτυσσόμενες χώρες χρειάζεται να στραφούν σε αγορές που έχουν ε, κανόνες πολύ πιο χαλαρούς. Συνεφώς δεν θα καταφέρουμε να επιρρήσουμε αυτό το πρόβλημα. Ξέρω ότι εκτιθέμεθα σε πολλές ομάδες πιέσεων, αλλά πραγματικά είχαμε καιρό να δούμε κάτι τόσο ανόητο σε αυτό που είδαμε σήμερα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συνάδελφο που θα ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Πραγματικά είναι ενδιαφέρον να μάθουμε πώς κατάφεραν οι άνθρωποι αυτοί να παρισφρήσουν στο Κοινοβούλιο. Ωραία, ας περάσουμε σε αυτά ε, προβλήματα. Εξυγίανση, ε, θέση σε διάθεση των δεδομένων. Στον τομέα των equities έχουμε συγκεκριμένες δομές που θα πρέπει να εξυγιανθούν και να αποκτήσουν έναν ευρωπαϊκό χαρακτήρα. Αυτό είναι η εξηγίαση των δεδομένων και αυτό θα, η ενοποίηση των δεδομένων και αυτό θα πρέπει να γίνει και για τα non-equities. Και εδώ υπάρχουν διάφορες τροπολογίες οι οποίες είναι υπέρ μιας μάλλον επιταχυμένης διαδικασίας. Αυτό για να επιτρέψουμε στους εποπτεύοντες οργανισμούς να παρεύουν σε διακρατικές σχέσεις. Αυτή είναι η πραγματική πρόκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Ηνωμένε Πολιτείε. Υπάρχει μία βασική, ένα βασικό χρηματιστήριο και ύστερα υπάρχουν τα περιφερειακά χρηματιστήρια. Εμείς έχουμε μεγάλα σημαντικά χρηματιστήρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για το λόγο αυτό είναι σημαντική η ενοποίηση των στοιχείων αλλά και ε, ο κανονισμός για την κατάχρηση των αγορών. Σε ό,τι αφορά τι ε, διακρατικές συναλλαγές έχουμε στη διάθεσή μας ε, λίγα δεδομένα. Σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα της corporate governance, τι, ε, ποια είναι τα προαπαιτούμενα εδώ για να μπορεί κανείς να διαχειριστεί ένα χρηματιστήριο. Περιμένουμε για να δούμε ποια θα είναι τα συστήματα ε, αυτά που θα επεξεργαστούν στο GED4. Θα πρέπει όμως να αποφύγουμε να τα κάνουμε όλα από την αρχή. Ήδη μιλήσαμε για αυτό το θέμα, χρειαζόμαστε ένα μέσο. Αρμοδιότητες του ΕΣΜΕ και αρμοδιότητες της Επιτροπής ακόμα και αν η Επιτροπή είναι εδώ παρούσα, θα πρέπει να πω ότι η πρόταση της Επιτροπής αναφέρει σε πολλά σημεία ότι τα προβλήματα θα πρέπει να λυθούν μέσω των πράξεων κατ' εξουσιοδότηση. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω προς ποια κατεύθυνση θέλουν να κινηθούν με αυτόν τον κανονισμό. Εγώ προτείνω μία συγκεκριμένη γραμμή που πιστεύω ότι την υποστηρίζουν οι συνάδελφοι και είναι η εξή. Εμείς ορίζουμε τον προσανατολισμό, προς τα πού θα κατευθυνθούμε. Όχι όμως μέσα από τις κατεξουσιοδότηση πράξεις, αλλά μέσω των προτύπων του ΕΣΜΑ όπου <clears throat> έχουμε το δικαίωμα τη αργή πράγμα που δεν συμβαίνει με τι κατεξουσιοδότηση πράξεις. Θέλουμε λοιπόν να ενισχύσουμε το ρόλο νομοθέτη. Και από την άλλη θέλουμε να έχουμε τη δυνατότητα να εκφράσουμε κάποια άποψη όταν τεθούν ορισμένα θέματα. Μη φύγει. Προτείνω να γίνει μια διάκριση μεταξύ των διμερών και των πολυμερών ε, συστημάτων. Γιατί όλες αυτές οι πλατφόρμες που υπάρχουν τα μύθη θα πρέπει να συμπεριληφθούν. Είναι, υπάρχουν πολυμεροί και υπάρχουν και διμεροί συστήματα, όπως είπαμε. Και αυτό θα πρέπει να οριστούν με, έναν όσο γίνεται ευρύτερο ορισμό. Έτσι ώστε ό,τι λαμβάνει η χώρα στον, εκτός μύθι να μπορεί να συμπεριληφθεί στον κανονισμό μύθιρ και Διαφάνεια. Πριν και μετά τη διαπραγμάτευση. Εδώ θα πρέπει να διευκρινίσουμε δύο σημεία. Καταρχάς το θέμα των commodities, των βασικών αγαθών και των παραγόγων. Πιστεύω ότι σε ό,τι αφορά την διαπραγμάτευση, ε, την διαφάνεια πριν από τη διαπραγμάτευση, υπάρχει ήδη μια καλή ρύθμιση, ένας καλός κανονισμός. Δεύτερον, στα πρέσια των κρατικών ομολόγων που τα πράγματα είναι διαφορετικά, Και εδώ υπάρχει διαφορετική ανάγκη για κανόνες διαφάνειας. Πιστεύω ότι αυτό είναι θεμητό γιατί η ομολογία είναι ένα ξεκάθαρο προϊόν. Οτιδήποτε επιλύεται μέσω του έμπειρ υπόκειται σε ένα σαφώς ορισμένο κανονισμό. Δεν θα πρέπει να δημιουργηθεί κάποιος κανονισμός ελέγχου σε ό,τι αφορά τα ό,τι σύστα χρηματιστηριακά προϊόντα. Όταν αυτά αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, αυτό θα πρέπει να λαμβάνει χώρα σε συγκεκριμένες πλατφόρμες, σε συγκεκριμένες χρηματιστηριακές αγορές. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να τίθεται υπό αμφισβήτηση το θέμα της πρόσβασης. Υπάρχουν βέβαια ορισμένε τεχνικές πτυχές που θα πρέπει να οριστούν καλύτερα. Τελευταίο σημείο, πάντοτε σε σχέση με το ΜΥΦΙ. Προτείνεται μια ευρεία απαγόρευση. Απαγόρευση ή περιορισμός για συγκεκριμένα προϊόντα, δραστηριότητες ή επιχειρήσεις. Πρόκειται για μια διάταξη εξ ας πούμε, ένας τίτλος θεωρείται ότι είναι αρνητικός, ότι είναι... Ε, ε κακός. εγώ θα έλεγα και εκ των προστέρων και εκ των υστέρων να, βρούμε. δρούμε. Κανένας βεβαίως δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για έναν ε, τίτλο, γιατί κάτι τέτοιο συνεπάγεται ε, κινδύνους. Συνεπώς το ΕΣΜΑ δεν μπορεί να βάλει τη σφραγίδα και να πει ότι συγκεκριμένη, ο συγκεκριμένος διαπραγματεύσιμος ε, τίτλος δεν έχει κινδύνους. Εκ των προτέρων όμως θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, δηλαδή να δούμε εάν το προϊόν αυτό συνεπάγεται ένα κίνδυνο. Στην περίπτωση αυτή η εποτεύουσα αρχή μπορούν, ναι, μπορεί να δράσει για να αποφευθούν οι αρνητικές επιπτώσεις. Ύστερα θα πρέπει να κάνουμε μία διάκριση μεταξύ για τα προϊόντα για τους ε, επαγγελματίες και για τους ε, πελάτες, για τους μικρούς ε, μετόχους. Εκεί θα μπορούσαμε να αυξήσουμε την προστασία του ε, καταναλωτή πολύ περισσότερο. Έλαβα 1140 τροπολογίες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους, του, όσους τις υπέβαλαν. Ήδη καταφέραμε να επιλύσουμε διάφορα προβλήματα. Θα κυκλοφορήσω, θα διανύμω προτάσεις συμβιβασμού. Προτάσεις οι οποίες θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Πραγματικά κατακλείστηκα από μηνύματα στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο. Γιατί υπάρχει ένα κανόνα ότι τίποτα δεν θεωρείται ότι έχει συμφωνηθεί αυτή τη στιγμή που θα συμφωνηθεί. Μέχρι στιγμή δεν έχει συμφωνηθεί τίποτα. Θα πρέπει να γίνει συζήτηση με του σκιώδει συζητητέ. Δεν υπάρχουν οριστικά κείμενα. Συνεπώ ελπίζω ότι θα μπορέσει να διατηρηθεί αυτή η επικοδομητική ατμόσφαιρα που χαρακτήρισε μέχρι στιγμή τι συζητήσει με του συναδέλφου. <clears throat> Αν θέλετε να έχουμε μια συζήτηση κατηδίαν, είστε πρόσδεκτοι στο γραφείο μου. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να δουλέψουμε με επικοδομητικό τρόπο για να σεβαστούμε τα χρονοδιαγράμματα και να τελειώσουμε πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Αυτό βέβαια δεν είναι κάτι που το λέω δογματικά. Γνωρίζουμε όμως ότι για έξι εβδομάδες δεν θα συναντηθούμε, δεν θα υπάρξουν συναντήσεις μεταξύ των σχεδόν εισηγητών. Θα ήθελα λοιπόν να είμαι έτοιμο πριν από το Συμβούλιο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μιλήσουμε τον Οκτώβριο για τη διαπραγματευτική εντολή. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι σημαντικό για τις ε, χρηματοπιστωτικές αγορές, ε, για τους πολίτες. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να περιοτώσει τις εργασίες του για να περάσει στη φάση των διαπραγματεύσεων. Ακύρωσα ορισμένες υποχρεώσεις που είχα στην εκλογική μου περιφέρεια ε, τις επόμενες εβδομάδες για να έχω χρόνο στη διάθεσή μου για να συζητήσω μαζί σας. Ελπίζω όλα να μπορέσουν να τελειώσουν μέσα σε ένα απόλυτα επικοδομητικό ε, κλίμα. Να καταλήξουμε σε ισχυρές και διαφανείς αγορές προς το συμφέρον όλων όσων συμμετέχουν σε αυτές τις αγορές. Ευχαριστώ. Thank you very much. I'll now move on to the Ευχαριστώ. Σαλή. Ευχαριστώ πολύ. And a very thoughtful uh, approach to the issue, which of course is complicated. It is an uh, extensive area that have. Ευχαριστούμε τον εισηγητή που έκανε αυτή την τόσο εμπεριστατωμένη εξήγηση στο θέμα αυτό, το οποίο είναι τόσο δύσκολο. Μιλώ εξ ονόματο του Ρόμπελ. Σε σχέση με λοιπόν την διαδικασία, ελπίζω ότι δεν θα καταδικάσουμε όλε τι ΜΚΟ για τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν και διαμαρτύρονται στη χώρα μου. Η Oxford και άλλες που αφορούν τα θέματα της πείνας έρχονται, μου στέλνουν email, μου μιλούν με τρόπο τον οποίο βρίσκω επικοδομητικό και χρήσιμο. Και όπως είπα δεν νομίζω ότι θα πρέπει να τους ε, καταδικάσουμε διότι ε, υιοθέτησαν αυτή την πιο επιθετική προσέγγιση που βεβαίως εγώ δεν ε, βρίσκω θετική. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρου του Ρόμπερτ που δεν παίρνω εδώ σήμερα, διότι είναι στη, με την αντιπροσωπεία μα στην Κύπρο, άρα δεν μπορούσε να συμμετάσχει στη συζήτηση. Όσον αφορά την ε, προσέγγιση. Ρόμπι, το θέμα αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Μάρκο και όλου του για την καλή του συνεργασία και για τι δύο επικοδομητικέ ήδη συναντήσει που είχαμε μέχρι τώρα. Πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί σε σημαντικές και επικοδομητικές τροπολογίες που θα βελτιώσουν την χρηματοπιστωτικές αγορές. Περιμένουμε τις ε, συνενετικές, να δούμε τι θα γίνει και ως οι συζητήσεις περιμένει να δει ποιες από αυτές θα περάσουν από αυτές που συζητήσουν. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό όλες οι χρηματοπιστικές επιχειρήσεις που ασχολούνται με αυτά τα θέματα, τα παράγωγα και τα σε ε, τέτοιου είδους συναλλαγές να προσπαθήσουν να ε, δίδουν τις ε, διαταγές και τις συναλλαγές τους να το κάνουν με ένα πλήρως διαφανές σύστημα και να μπορέσουν να μας δίνουν όλες τις πληροφορίες για να μπορούν οι υπεύθυνοι να μπορέσουν να κάνουν την κατάλληλη εποπτεία του τι ακριβώς γίνεται. Επίσης, θα πρέπει να δούμε τι ε, γίνεται με το θέμα αυτών των συναλλαγών των αλγοριθμικών της υψηλής συχνότητας. Νομίζω ότι θα πρέπει να συστήσουμε μία συμβουλευτική ομάδα για το θέμα αυτό των συναλλαγών υψηλής συχνότητας. Επίσης, για τη δομή της αγοράς, στα πλαίσια των ε, κανονιστικών ε, δομών που έχουμε, θα πρέπει να έχουμε ένα ε, πλαίσιο για το trading, για όλες αυτές τις συναλλαγές. Θα πρέπει όπου υπάρχουν ε, ε, αδυναμίες και προβλήματα στον κανονισμό να μπορέσουμε να τα ρυθμίσουμε ώστε να μην προκαλούμε προβλήματα στην αγορά, να βελτιώσουμε την δυνατότητα των ρυθμιστικών αρχών να εποπτεύω την αγορά και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνουν κάποιες διορθώσεις ώστε να μην προστρέχουν και κάποιοι σε κακή ερμηνεία του κανονισμού ε, μη Επίσης θα πρέπει να δούμε τις πολυμερείς και διμερείς συναλλαγές. γίνεται παράκληση στην ομιλήτρια που διαβάζει ένα κείμενο για ένα τόσο πολύπλοκο θέμα που δεν έχουν οι διερμηνείς να μιλά λίγο πιο αργά. Ευχαριστούμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι για κάποιους δεστρέχουσες συναλλαγές της αγοράς θα πρέπει να δούμε πώς θα ρυθμίσουμε διάφορα ε, προβλήματα όπως ε, αυτό των έξω χρηματιστηριακών συναλλαγών, των OTCs, στα πλαίσια των αγορών. Και πώς θα μπορέσουν να γίνονται κάποιες συναλλαγές, οι όλες οι συναλλαγές με ασφάλεια. Υποστηρίζουμε την έκθεση η οποία έγινε το Dark Pools που επίσης ψηφίστηκε στην Ολομέλεια ώστε να υπάρχουν και νέοι τόποι trading. Οι πολυμερείς μηχανισμοί διαπραγμάτευσης επίσης θα πρέπει να, γι, να έχουν διαφάνεια και να μην υπάρχουν διακρίσεις όσον αφορά την εποπτεία των αγορών ή τα αντικρουόμενα συμφέροντα, ώστε όλες οι συναλλαγές να γίνονται με ασφάλεια. Όσον αφορά το ότι εύτης πολυμερούς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ώστε να μην ε, υπάρχει σύγχυση και οι διάφοροι ιδιωτικοί επενδυτές να γνωρίζουν πολύ καλά σε ποια πλαίσια κινούνται. Επίσης, οι πολυμερείς μηχανισμοί διαπραγμάτευσης θα πρέπει να περιοριστούν στο non-trading equities και να μπορέσουμε να θεσπίσουμε κανόνες που να βοηθήσουν την αγορά να κινείται με ασφάλεια. Επίσης, θα πρέπει να δώσουμε σαφή ορισμό στο θέμα αυτό των έξω χρηματιστηριακών συναλλαγών, των over-the-counter transactions. Θα πρέπει να έχουμε σαφή μέτρα, σαφείς κανονισμούς και να μην δημιουργήσουμε σύγχυση στις αγορές. Ο κατακαιρματισμός των αγορών ξέρουμε ότι δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στην εποπτεία τους και θα πρέπει να προσέξουμε τα παραθυράκια. Ξέρουμε ότι με τις τροπολογίες που καταθέτουμε θα πρέπει οι εξοχρηματιστηριακές συναλλαγές να γίνουν πιο ασφαλείς Όσον αφορά το SED, τα Position Management, δεν θα πρέπει να το ενθαρρύνουμε. Οι διάφορες αρχές θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες που να αφορούν και τους συλλογικούς και τους μεγάλους και τους μικρούς ιδιωτικούς επενδυτές ώστε να ξέρει κανείς ποιες είναι οι ασφαλείς συναλλαγές κυρίως στον εμπορικό κόσμο. Τώρα, ε πρώτες ύλες ξέρουμε ότι επηρεάζονται και από άλλα θέματα. Θα πρέπει να ισχύουν στις αγορές οι αρχές της αμοιβαιότητας και της ισοδυναμίας για την προστασία των καταναλωτών πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν σαφείς κανόνες για τους διαμεσολαβητές ώστε να υπάρχει, να, ε, για να ισχύει για όλους να ισχύουν για όλους οι ίδιοι κανόνες δεοντολογίας και να προσάγονται και στη δικαιοσύνη αυτοί οι οποίοι δεν ενεργούν με σωστό τρόπο. Τα άρθρα 28 και 29 στον κανονισμό η Επιτροπή προβλέπει τι γίνεται σε περίπτωση μη αποτελεσματικότητας ή δυσλειτουργία στην αγορά που μπορεί να δημιουργήσει ακόμη περαιτέρω κατακαιρματισμό. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε το σύστημα που λειτουργεί σωστά να συνεχίσουμε να το υποστηρίζουμε και να μην το αφήσουμε να υποκατασταθεί από αυτούς που θέλουν να καταχραστούν τους κανόνες, τους σωστούς κανόνες στην αγορά. Θα πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός υγιής στην αγορά και να μπορούμε να βοηθούμε και να προστατεύουμε τους επενδυτές. Κυρίως για τα έξω χρηματιστηριακές συναλλαγές και τα παράγωγα, χωρίς διακρίσεις. Η αγορά ήδη κατακαιρματισμένη. Ξέρουμε ότι, δημιουργεί, ότι έχει προβλήματα και θα πρέπει όποια ρύθμιση να γίνει με τρόπο που να έχουν όλοι ε, την ίδια ε, πρόσβαση και οι κανόνες που θα λειτουργούν στις ε, μη ρυθμιζόμενες αγορές να είναι οι ίδιοι με αυτούς που ισχύουν για τις ρυθμιζόμενες αγορές. Θέλουμε να δημιουργήσουμε σταθερότητα στην αγορά στο άρθρο 29 νομίζω ότι εντείνεται ο κατακαιρματισμός των αγορών. Θα πρέπει λοιπόν να μην επιτρέψουμε κάτι τέτοιο, διότι οι αγορές πραγματικά θα είναι εφιάλτης για όλους. Τελειώνοντας, ε, ήθελα να πω ότι ο κύριος Γκέμπελς θέλει να συνεργαστεί με τον κύριο Φέρμπερ για να μπορέσουν να καταλήξουν σε συμβαστικές τροπολογίες. Ευχαριστώ. Όλε Σμιτ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομος γίνεται, διότι νομίζω ότι αυτά τα επιχειρήματα τα είχα αναφέρει και την προηγούμενη φορά. Αρχίζοντας πρέπει να πω ότι νομίζω ότι κάνει εξαιρετική δουλειά ο Μάρκους Φέρμπερ. Έχετε δει όλοι τις συμβιβαστικές τροπολογίες, τα έχουν δει δηλαδή και οι διάφορες οργανώσεις, οι ε, Άρα νομίζω ότι είναι γνωστές και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ευρεία συνέντευξη. Πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό, λαμβάνοντας υπόψη την ε, κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται σήμερα. Μπορώ να το διαβλέψω. Φαντάζομαι ότι μπορούμε να το κατορθώσουμε κάτι τέτοιο. Και μου αρέσει που το λέω. Τώρα, όσον αφορά αυτή την ε, δια, μικροδιαδήλωση που έγινε εγώ. Εμένα είμαι μέλος της Επιτροπής για την Αφρική. Και ήμουν πέρσι στη Ζάμπια. Σήμερα η Ζάμπια είναι μία από τις πιο φτωχές χώρες του κόσμου. Και τι κάνει στην περιοχή της εξάγει αγροτικά προϊόντα. Υπάρχουν λοιπόν κάποια μηνύματα ελπίδας και θα ήθελα να πω ότι το πιο σημαντικό για να μπορεί κανείς να παρέχει Ήδη διατροφής με ασφάλεια στην Αφρική να δημιουργήσει ε, μία αγορά με ευαισθησία, πράγμα το οποίο δεν θα πρέπει η ΚΑΠ στην Ευρώπη να καταστρέψει. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό και θα πρέπει να το πούμε. Έξι θέματα με απασχολούν, κυρία Πρόεδρε, τα οποία θα ήθελα να σας τονίσω. Τα OTF καταρχά. Νομίζω ότι τα OTF τα χρειαζόμαστε. Είμαι υπέρ αυτής της ε, κατηγορίας όπως συμβαίνει και με τα μετοχικά προϊόντα. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μεγαλύτερη διαφάνεια και μεγαλύτερος ανταγωνισμό για όλα τα μέσα. Χρησιμοποιείται ένα, δημιουργείται ένα πεδίο αμβλύνονται οι διαφορές και βεβαίως είναι σύμφωνο, είναι ευθυγραμμισμένο με τις δεσμεύσεις που έχουν αναλυφθεί στη συνάντηση των ε, G12. Μιλάμε πάντοτε για τους πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης. Για μένα αυτό είναι σημαντικό, είναι κάτι που θα πρέπει να τονίσουμε. Παρέχει και μια ελευθερία επιλογών η απαγόρευση σε ένα χειριστή ότι να μην χρησιμοποιήσει το κεφάλαιό του, κατά την άποψή μου είναι ιδιαίτερα αυστηρό και ενδεχομένως περιορίζει τη δυνατότητα να παρέχουμε την καλύτερη δυνατότητα εκτέλεση στους πελάτες μας. Συμπερασματικά θα έλεγα ότι είμαι υπέρ μίας μορφής OTF. Καταλαβαίνω ότι ο Μάρκους κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να ορίσει το πώς, την εικόνα που θα έχει αυτός ο περιμερής μηχανισμός διαπραγμάτευσης. Εμείς όμως θα μπορέσουμε να επιτύχουμε ένα συμβιβασμό. Διαφάνεια. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό το να επιτευχθεί μεγαλύτερη διαφάνεια και καλύτεροι κανόνες διαφάνειας. Ανέφερα την προηγούμενη φορά που πήρα το λόγο ότι έχω κάποιο προβληματισμό. Και αυτό το Παρέφερε και ο Μάρκους ότι δεν είναι τόσο εύκολο να υπάρξει διαφάνεια πριν από την διαπραγμάτευση. Θα πρέπει να υπάρχει εξισορρόπηση από την ανάγκη να ε, ε, ε, δημιουργηθούν προβλήματα στην αγορά. Αναφέρθηκε βεβαίω και το θέμα των κρατικών ομολόγων, της αγοράς των κρατικών ομολόγων. Νομίζω ότι μέσω των προτάσεων συμβιβασμού θα μπορούσε να επιτευχθεί ένα συμβιβασμό και σε ό,τι αφορά αυτό το σημείο. Δεν χρειάζεται να αναφερθώ εκτενέστερα σε αυτό το θέμα. Ελπίζω να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε ε, εκ δεξιών ή μάλλον εξ αριστερών καθήμενος φίλος μου ελπίζω να συμφωνήσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Μάρκους είπε πολλές φορές ότι δεν χρειαζόμαστε περισσότερα προβλήματα σε ό,τι αφορά την αγορά των ομολόγων στην Ευρώπη. Αρκετά προβλήματα είχαμε μέχρι τώρα. Προστασία των επενδυτών. Και εκεί διαπιστώνω ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί μια συμφωνία. Ε, συνένεση, συμφωνώ με την πρόταση του Μάρκους να στοχεύσουμε συγκεκριμένα προϊόντα σε συγκεκριμένους πελάτες και να μην υπάρχει πλέον η έννοια της ανεξάρτητης συμβουλής. Γιατί δεν είναι δυνατόν να υπάρχει μια τέτοια συμφωνία μεταξύ των διαμεσολαβητών και των τραπεζών γιατί και εδώ θα μπορούσαμε να δούμε ότι έχουμε διατυπωθεί ορισμένες λογικές προτάσεις. Αναφέρθηκε στο θέμα της επικουρικότητας ή μάλλον χρησιμοποίησε μια άλλη λέξη, μια γερμανική έκφραση. Είχα την εντύπωση ότι προερχόταν από μια ταινία με τον Σον Κόνερι. Εντάξει, εντάξει. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε λίγο περιοριστικοί στον τομέα αυτό. Η αλγοριθμική διαπραγμάτευση, διαπραγμάτευση ψηλής συχνότητας. Βεβαίως υπάρχει αυτή η ιστορία με τα FTT και όλα αυτά. Χρειαζόμαστε κάποια πολιτικά σύμβολα. Συμφωνώ. Πιστεύω ότι το FTT είναι μια πραγματικότητα και ενδεχομένω ε, να χρειαζόμαστε και κάτι άλλο. Ενδεχομένω θα μπορούσαμε να το δούμε εκτενέστερα το σημείο αυτό στο κείμενο. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να το διατυπώσουμε κάπως καλά. Ο Μάρκους έχει ορισμένες προτάσεις σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις και νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε μία ε, διαφοροποίηση μεταξύ του ε, HFT και του, ε, και της διαπραγμάτευσης του algo trading. Εδώ έχουμε ένα άλλο θέμα που θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε κάποια συζήτηση. Αυτά το 500 milliseconds αν, αν προτείνω 500 ή 400 μιλισέκοντς, αυτό θα σας έβρισκε σύμφωνους. Δεν ξέρω. Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε μία άλλη μέθοδο. Και είδα ότι ορισμένοι συνάδελφοι αναφέρθηκαν σε πέντε δεύτερα. Μιλάνε για ένα διάστημα δύο ετών κατά τη δική τους άποψη. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε κάποιο άλλο σύστημα. Δεν ξέρω, συγκεκριμένους κανόνες ενδεχομένως. Βεβαίως καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι τεχνικό πρόβλημα, θα μπορούσε να είναι πρόβλημα της αγοράς και ενδεχομένως και πολιτικό πρόβλημα. Συμφωνώ με αυτό. Πρόσβαση στις υποδομές της αγοράς. Ελπίζω ότι και εκεί θα μπορούσαμε να επιτύχουμε μια συμφωνία. Πρόκειται για ένα ευαίσθητο θέμα. Όλα αυτά τα θέματα είναι ευαίσθητα βέβαια. Εγώ είμαι υπέρ της δίκαιας και ε, ανοιχτής πρόσβασης στα CCP. Αυτό είναι σημαντικό να μην, ε, για να μην δημιουργηθεί μια συγκέντρωση των κινδύνων. Βεβαίως ε, χρειάζεται ο ανταγωνισμός. Και αντί να επικεντρώσουμε την αγορά, θα επιτρέψουμε και σε άλλες συσυπείς να παράσχουν τις υπηρεσίες τους. Αυτό θα οδηγήσει σε περισσότερες ε, καινοτομίες. Αυτό είναι ένα από τα σημαντικά θέματα εδώ. Δεν θα πρέπει να περι, τα περιορίσουμε όλα αυτά μιλώντας για τους τόπους διαπραγμάτευσης σε κεντρικούς αντισυμβαλόμενους για τα CCPs. Υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο. Υπάρχει, χρειάζεται ένας καλύτερος καταμερισμός κινδύνου μεταξύ αυτών των τόπων διαπραγμάτευσης. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για ένα πραγματικό συστημικό κίνδυνο. Τέλος, τρίτη χώρα. Συμφωνώ με αυτό που είπε ο Μάρκος. Πολλοί από εμά εδώ, η πλειοψηφία, δεν έχουμε τα αγγλικά ως αμυτρική μας γλώσσα και χρησιμοποιούμε αυτά τα κουτσά αγγλικά. Τώρα, ποια είναι η διαφορά μεταξύ ισοδυναμίας και αμοιβαιότητας. Για μένα αμοιβαιότητα ρεσιπρόσιτη χρησιμοποιείται πάντοτε ως πολιτικό σύμβολο για τα ε, για τη δημιουργία προσκομμάτων. Εγώ έτσι την ερμηνεύω την αμοιβαιότητα. Συνεπώς είμαι υπέρ της χρήσης του όρου ισοδυναμία. Και αν αυτό σημαίνει ότι αυτοί που θέλουν να προωθήσουν την ιδέα της ε, αμοιβαιότητας. Αυτό θα καταστήσει περισσότερο δύσκολες τις επενδύσεις στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Θα έλεγα ότι είμαι αναφανδόν κατά και νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ κακό και αυτή την Επιτροπή το να προσπαθήσει να καταστήσει πιο δύσκολες επενδύσεις στην Ευρώπη αυτές τις μέρες. Για δέστε τι γίνεται σήμερα στο Μεξικό. Όλοι έχουν στραμμένα τα μάτια στην Ευρώπη και η Ευρώπη λέει ότι δεν φταίμε εμείς. Μπορούμε να τα πάμε καλύτερα και χρειαζόμαστε επενδύσει, χρειαζόμαστε χρήματα απ' έξω. Θα πρέπει λοιπόν να μας ε, οδηγήσουν σε σκέψεις όλα αυτά. Πραγματικά με βρίσκει σύμφωνος ο τρόπος με τον οποίο διαδραμάτισες το ρόλο σου ως εισηγητή σε ένα πολύ ευαίσθητο θέμα και στα πλαίσια της ομάδας Άλτη θα κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να επιτευχθεί μια συμφωνία. Θα σταματήσω εδώ γιατί βλέπω ότι υπάρχουν συνάδελφοι που θέλουν και εκείνοι να αναφερθούν σε αυτό το θέμα. Στην ομάδα μας πραγματικά καταβάλαμε προσπάθεια στο να καταλήξουμε σε ένα λογικό συμβιβασμό. Ενδεχομένως το φτάσαμε, αλλά θα ήταν χρήσιμο να γίνουν και μερικά επιπλέον σχόλια. Ευχαριστώ πολύ. Μετά έχουμε τους ε, πράσινους στην λίστα μας. Υπάρχει πάντα αυτή η συζήτηση, αλλά τέλος πάντων η πράσινη πράσινοι επόμενοι. Σφέν. Και εγώ έχω συγχυστεί λίγο για, σε σχέση με τους κανόνες. Έχω μια σύγχυση. Ε, συνήθως είμαστε σε μικρότερο κλίμακα στην Επιτροπή μας, τώρα είμαστε σε μεγαλύτερη κλίμακα εδώ στην Ολομέλεια. Ίσως πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, αλλά δεν είναι και το πιο ε, σημαντικό θέμα στον κόσμο, ποιος μιλάει πρώτος. Ας ε, συμφωνήσουμε γι' αυτό. Λοιπόν, από την πλευρά μου ευχαριστώ τους εισηγητές ε, για, την καλή, για τον εισηγητή για την καλή συνεργασία. Ε, πάντοτε ήσασταν διαθέσιμος όποτε ζητήσαμε να σας δούμε. Αυτό ε, με χαροποιεί. Μετά ε, υπάρχουν κάποια άλλα θέματα ε, που θέλω να θίξω. Να πω ότι ο Σκιώδης Πασκάλ Κομφάν είναι τώρα Υπουργός Ανάπτυξης ε, και αν ε, καταλαβαίνω σωστά τη γαλλική πολιτική που πραγματικά δεν την καταλαβαίνω βλέποντας κάποιες από τις πρόσφατες αποφάσεις τους, τέλος πάντων αν καταλαβαίνω σωστά ο Πασκάλ ε, θα παραμείνει στη θέση του, οπότε δυστυχώς δεν θα συνεχίσει εδώ, το οποίο έχει και το αρνητικό αποτέλεσμα ότι πρέπει να αναλάβω αυτό το πολύπλοκο έγγραφο με τις 2.000 και τόσες τροπολογίες τελευταία στιγμή. Ε, αν δούμε το τεράστιο πεδίο της ΜΥΦΙΤ, βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα που εγείρονται ε, σχετικά με το αν είναι χρήσιμη αυτή η οδηγία ως μια μεγάλη οδηγία. Είναι κάτι που πραγματικά πρέπει να συζητηθεί. Έχοντας ε, ε, δει πόσο λίγο χρονικό περιθώριο υπάρχει για συμβεβασμούς σε τόσο πολύπλοκα θέματα, ε, καταλαβαίνω ότι μπορεί να υπάρξουν δυσκολίες να γίνει κάτι τέτοιο μέχρι το καλοκαίρι. Και πραγματικά προσυπογράφω αυτό που είπε ο Μάρκος Φέμπερ, ότι θα προσπαθήσουμε σκληρά να υπάρξει συμβιβασμός, ο, η συνένεση μάλλον, αλλά αυτό θα έχει το αρνητικό ότι δεν θα υπάρχουν ε, συζητήσεις εις βάθος ε, και κάποια από τα ζητήματα είναι πολύ τεχνικά. Όπως υπόθηκε, πολλές φορές ε, μπορεί τεχνικά ε, να κάνουμε κάτι λάθος με διαφορετική πρόθεση και στο τέλος να πετύχουμε το αντίθετο από αυτό που θέλουμε. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει ε, να είμαστε πολύ συνειδητοποιημένοι ως προς το τι κάνουμε εδώ. Τώρα, για τα διάφορα θέματα που μας αφορούν. Ε, πολλά υπόθηκαν για το θέμα των οργανωμένων μηχανισμών διαπραγμάτευσης, τα OTFs. Εγώ να πω ότι αυτός ο νέος μηχανισμός ε, ε, θα πρέπει να παραμείνει σε πολύ στενά όρια στα μη μετοχικά προϊόντα και στους ε, επαγγελματίε επενδυτές. Νομίζω ότι αυτό είναι κοντά σε αυτό που προτείνει ο εισηγητής. Υπάρχει λόγος να υπάρχουν αυτοί οι μηχανισμοί και υπάρχει κίνδυνος αν δεν υπάρχουν τέτοιοι κανόνες γιατί στο τέλος θα έχουμε όλο και περισσότερες ε, ε, τρύπες, όλο και περισσότερα κενά, ε, παραθυράκια και χώρους αριθμιστούς, πεδία αρρύθμιστα και γι' αυτό ας μην είμαστε πολύ φιλελεύθεροι και να αφήσουμε αυτά τα περιθώρια. Να πω λοιπόν ότι σωστό είναι που μπαίνει αυτή η νέα κατηγορία, αλλά να υπάρχουν πολύ αυστηροί κανόνες γι' αυτό. Μετά υπάρχει το θέμα των παραγόγων. Ε, σύμφωνα με, την, ε, με τον Εμμύρ, ήδη ήταν δύσκολο να ε, οριστούν ε, τα τυποποιημένα παράγωγα ε, που έχει να κάνει με τους μακρο πρόθεσμους χρήστες, ε, του hedges και όλους αυτούς που χρησιμοποιούν αυτά τα παράγωγα. Ε, στο MIFID ε, καλύπτονται όλα αυτά τα παράγωγα που χρησιμοποιούνται για clearing. Έτσι λοιπόν, όπως έχουν πει και πολλοί ευρωβουλευτές, υπάρχει αυτό το ζήτημα πολύ σημαντικό. Πρέπει επίσης να λαμβάνουμε υπόψη μας ότι η απουσία ρευστότητα σε ένα προϊόν δεν θα ε, πρέπει να αποτελεί λόγο άρσης ε, της, ε, των υποχρεώσεων. Αν ένα τυποποιημένο προϊόν βρίσκεται εκτός του ΕΜΗΡ σε πλατφόρμα MIFID, θεωρούμε ότι θα πρέπει και πάλι να υπάρχει υποχρέωση διαπραγμάτευσης σε ρυθμισμένο τόπο, έτσι ώστε να αποφευχθεί η συνύπαρξη ε, εξοχρηματιστριακών ε, κύκλων ε, και τέτοιων προϊόντων για να πετύχουμε τους στόχους του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Θα πρέπει λοιπόν να πάμε στα πιο τυποποιημένα προϊόντα, σε πιο ε, συγκεκριμένους τόπους, πιο ρυθμισμένους τρόπους. Ε, οι συναλλαγές ε, οι εξοχρηματιστηριακές ε, θα πρέπει να περιορίζονται σε πολύ συγκεκριμένα παράγωγα που χρησιμοποιούν στις συναλλαγές τους οι επαγγελματίες επενδυτές και οι εταιρείες επενδύσεων. Έτσι, καλωσορίζω τα ε, σχόλια των συναδέλφων από τις άλλες ομάδες ε, είπατε ας πούμε ότι ε, πρέπει να υπάρχει κάποιος ορισμός για όλα αυτά. Να πω επίσης κάποια πράγματα για την προστασία των καταναλωτών. Καταρχάς, υποστηρίζουμε τη βασική προσέγγιση του εισηγητή να εισαχθούν διάφορες τάξεις προϊόντων που μπορεί να μην είναι κατάλληλα για retail, για λιανική πώληση, και και που δεν έχουν επιπλέον αξία για τους ε, καταναλωτές. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει ε, μία εκ των προτέρων ε, παρέμβαση για κάποια τέτοια προϊόντα. Πέρα από αυτό, σε αυτό το πεδίο βλέπουμε κάποια πολύ σημαντικά ζητήματα για τους καταναλωτές και τους ανθρώπους που είναι πελάτες λιανικής, οι οποίοι χρειάζονται και αξίζουν αυτή την προστασία προσφέρονται συμβουλές, όμως δεν είναι αυτό που συνήθως ε, λέμε ε, παροχή συμβουλών. Ε, συνήθως ο σύμβουλος είναι με την πλευρά σου. Όμως εδώ έχουμε μία διαδικασία πώλησης και στις πωλήσει αυτό θα πρέπει να ονομάζεται προσπάθεια πώλησης και όχι παροχή συμβουλών. Έτσι λοιπόν ε, οι συνάδελφοι Καμάλ και Σουίνμπορκ προτείνουν τροπολογίε σχετικά με τη συμπερίληψη ενός ορισμού για τις ε, επενδυτικές υπηρεσίε που βασίζονται ε, σε ασφαλιστικά προϊόντα. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τους καταναλωτές να συγκρίνουν διάφορα προϊόντα. Επίσης, κατέθεσαν άλλες τροπολογίες, τις οποίες προσπογράφουμε, αποκάλυψη κόστου επενδυτικού είναι λίγο πολύ στη γραμμή αυτού που προτείνουμε κι εμείς. Εμείς θεωρούμε ότι η απαγόρευση για, ε, των προμηθειών για ανεξάρτητες συμβουλές ε, καλύπτει μόνο ε, μέρος του προβλήματος. Σύμφωνα με τη Βρετανική εμπειρία, λοιπόν, η Κομισιόν προτείνει κάτι που δεν αγγίζει τον ευρύτερο χώρο των πελατών λιανικής που είναι οι τράπεζες και γι' αυτό ε, το να απαγορεύουμε ε, από τις τράπεζες την ανεξάρτητη συμβουλή, ε, τότε απλώς διαγράφει το όρος ανεξάρτητος και συνεχίζουν τα πράγματα όπως πριν. Ε, ίσως, αν περάσουν οι συναλλαγές στην τράπεζα και σε ομάδες, θα μειωθεί ο ανταγωνισμός. Στο τέλος, θα έχουμε δεν θα έχουμε περισσότερη διαφάνεια και ε, σύγκρουση, λιγότερη σύγκρουση συμφερόντων, αλλά περισσότερη συγκέντρωση. Γι' αυτό θεωρώ ότι τα κίνητρα που δίνονται στους συμβούλους θα πρέπει να δίνονται ε, πλήρως στους καταναλωτές ώστε να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων ε, για την παροχή συμβουλών για το προϊόν Α ή Β μόνο και μόνο επειδή έχει περισσότερα κίνητρα. Αυτό έχει να κάνει με τους ανεξάρτητους συμβούλους ε, και την παροχή αδέκαστων συμβουλών. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, δεν μας αρέσουν οι τροπολογίες που κατατέθηκαν για να απαγορεύσουν στα κράτη-μέλη να έχουν μια ε, προνοητική ας πούμε προσέγγιση ε, απαγορεύοντας την κατάργηση των κινήτρων για τους ανεξάρτητους συμβούλους. Έτσι λοιπόν η Ευρώπη λίγο πολύ με αυτόν τον τρόπο ε, παρεμβαίνει κατά κρατών μελών που έχουν λίγο πιο εκτεταμένους κανόνες. Έχουμε επίσης ε, τροπολογίες από λίγο πολύ όλες τις ομάδες για την εισαγωγή μεγαλύτερων, ισχυρότερων μάλλον τεστ καταλληλότητας. Εμείς έχουμε σοβαρές αμφιβολίες ε, ότι αυτό θα είναι δικαιολογία για να εξαιρεθεί η χρήση από το πεδίο των κανόνων MIFID. Θεωρούμε επίσης ότι οι συμβουλές για τη χρήση θα πρέπει να περιλαμβάνεται ε, στο πεδίο το, της προστασίας των καταναλωτών. Επίσης, να κλείσω με κάτι άλλο που, υπήρχε και, που έγινε και ο λόγος για αυτή την διαμαρτυρία. Να πω ότι Υπάρχουν κάποιες εκδηλώσεις για τις χρηματοπιστωτικές αγορές στη Γερμανία, ε, στις οποίες πραγματικά ε, αυτό που φαίνεται ότι αγγίζει τον κόσμο περισσότερο είναι η κερδοσκοπία με το φαγητό. Άρα είναι ένα βαθύ ηθικό πρόβλημα και γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ ε, προσεκτικοί στο πόσο εκρίνουμε τις παρεμβάσεις από το κοινό. Υπάρχουν πολλές προτάσεις, πολλά άρθρα, αλλά όπως είπε η Άλλη Μακάρθη, γι' αυτό το θέμα έχουμε τους μεγάλους αναπτυξιακούς οργανισμούς, αυτούς ε, που σχετίζονται με την Εκκλησία Oldford, Die Welt, Miseria και άλλες όπως η Oxfam, που όλες ε, αυτές οι οργανώσεις ανησυχούν και παρακολουθούν στενά τι κάνουμε. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί, να μην κρίνουμε λανθασμένα οποιαδήποτε μορφή δημόσια δραστηριότητα. Ακόμα και η δημοκρατία μπορεί να αντέξει μερικά ε, δευτερόλεπτα διακοπής των εργασιών, ακόμα και σε αυτό την αίθουσα της Ολομέλειας. Ε, για ε, τους πόρους τώρα που, χρησιμοποιούνται τα, που χρησιμοποιούν τα λόμπι ε, κερδοσκοπίας, ε, καταλαβαίνετε ότι έχουμε μια ανοχή. Γιατί λοιπόν όχι σε αυτό. Ε, υπήρξε πολύ μεγάλη αναστάτωση ως προς αυτό που είδαμε εδώ μέσα. Ε, σε σύγκριση με το τι γίνεται κάθε μέρα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία κάθε μέρα ε, εκτοξεύουν δεξιά και αριστερά μηνύματα σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές αγορές και το τι πρέπει να γίνει. Θα πρέπει να προσέχουμε, αλλά και θα πρέπει να χαιρόμαστε που κάποιοι παρακολουθούν στενά το τι κάνουμε με, με κριτικό πνεύμα. Αυτά είχα να πω. Ε, προσβλέπω στη συνεργασία με τους συναδέλφους για αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Και τώρα για το ECRK. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να ξεκινήσω ευχαριστώντας ε, τον εισηγητή για την πρόοδο που, είχε, που έχει καταφέρει ήδη σε ένα τόσο μεγάλο θέμα σήμερα. Υπάρχει πρόοδο σε πολλούς τομείς. Οι απόψει μου είναι πολύ γνωστές στα περισσότερα από τα θέματα των υποδομών της αγοράς, ε, γιατί παρακολουθώ στενά τις εργασίες. Υπάρχουν κάποια θέματα που θέλω τώρα να θίξω σήμερα που έχουν όλα να κάνουν με τον ανταγωνισμό. Η πρόσβαση, η συζήτηση για τις αγορές μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τρίτον ε, το καθεστώς των ε, τρίτων χωρών. Στην αρχική και ο στόχος ήταν η αύξηση του ανταγωνισμού ειδικότερα στις αγορές μετοχικών προϊόντων, δημιουργώντας μια ε, υποδομή της αγοράς και αφαιρώντας τους κανόνες συγκέντρωσης. Ήδη έχουμε αλλάξει το περιβάλλον των συναλλαγών με τη MIFID 1. Τώρα θέλουμε να έχουμε και πάλι αυτό το στόχο του θετικού ανταγωνισμού ε, στην ε, στις υποδομές ε, που τώρα θα ρυθμίσουμε. Έχω προσωπικά λίγες τροπολογίες για τα άρθρα 28, 29 και 30 στο κείμενο της Κομισιόν. Θεωρώ ότι σωστό σωστά χρησιμοποιεί η Κομισιόν αυτή τη ρύθμιση της αγοράς ε, για να ε, φτάσουμε σε μια πιο ανταγωνιστική αγορά. Αν μπορούμε να φτιάξουμε ένα νομοθέτημα ε, σωστό για την αγορά ελέγχου ε, και της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας πριν από χρόνια, αν τα είχαμε καταφέρει, ε, Τώρα δεν θα είχαμε αυτό το πρόβλημα με κάποιους παίχτες που έχουν υπερβολική ισχύ και παρέχουν υπηρεσίες στην Ευρώπη. Υπάρχουν συζητήσεις για το πώς μπορεί να αφαιρεθεί αυτή η δυνατότητα κυριαρχίας στην αγορά. Ε, πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να διαγραφούν αυτά τα άρθρα που διασφαλίζουν ε, τον ανταγωνισμό. Ε, αυτοί οι Ευρωπαίοι ε, πρωταθλητές ε, για μένα δεν είναι κάτι που κατανοώ. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ώστε τα θεσμικά όργανα που διαθέτουμε να είναι τα καλύτερα δυνατά ε, και να μπορούν ε, να βοηθούν τις, τα κράτη να καινοτομούν και να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες στην αγορά. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ανοιχτή μη, ε, πρόσβαση χωρίς διακρίσεις σε όλες τις υποδομές και θα πρέπει αυτό να το καλωσορίζουμε ως στόχο ανταγωνισμού για όλες τους θεσμούς. Τώρα για τα ε, αγορές ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έχω τροπολογίες δεν έκανα τροπολογίε στο άρθρο 35 της Κομισιόν γιατί θεώρησα ότι ε, πάει στη σωστή κατεύθυνση. Η αποδοχή μιας διαφορετικής τάξης ε, η οποία ε, αναγνωρίζεται ως αγορά ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε τη δυνατότητα στο μέλλον να έχουμε νομοθετικές προτάσεις ε, οι οποίες θα τις αντιμετωπίζουν χωριστά. Έτσι στην ε, οδηγία ας πούμε διαφάνειας ε, ή προοπτικών του νόμου ασφάλειας αυτό θα μας βοηθήσει. Η νέα κατηγορία της MIFID θα βοηθήσει να, αν κάποιο κράτος μέλος θέλει να ενισχύσει την ανάπτυξη μέσα από αυτό το τομέα, να έχει τα κατάλληλα εργαλεία. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτή την ε, ξεχωριστή κατηγορία και να έχουμε σωστό ορισμό της, έτσι ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορέσουν να αναπτυχθούν ε, γρήγορα και σωστά και να είναι έτοιμοι να ε, μπουν στην κύρια αγορά στο άρθρο 4 παράγραφος 2 σημείο 12 η Κομισιόν προσπάθησε να δώσει μια τυπική, ένα τυπικό ορισμό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, μιλάει εκεί και για τις ε, κρατικές ενισχύσεις, όμως αυτό δεν ε, έχει να κάνει με το τι είναι η αγορά ανάπτυξης. Συνεπώς ε, θα ήθελα να ζητήσω έναν ορισμό που να συμπεριλαμβάνει την επανακεφαλοποίηση της αγοράς όχι μόνο τον αριθμό των εργαζομένων και τον κύκλο εργασιών. Ξέρω ότι καταρχάς συμφωνεί ο εισηγητής με την ανάπτυξη αυτής της κατηγορίας και ελπίζω ότι ένα συμβιβασμό θα βοηθήσει αυτή την ομάδα να προχωρήσει. Δεν θέλω να, προσ... περάσω στο θέμα των τρίτων χωρών. Ο ίδιος ο εισηγητής το ανέφερε, το ανέφερε και ο κύριος Σμιτ στα σχόλιά του. Πραγματικά δεν θέλουμε οι αγορές της Ευρώπης να βάζουν προσκόμματα στους επενδυτές και δεν θέλουμε να περιορίσουμε τις εισρωές κεφαλαίου εκτός και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκείνο που θα πρέπει να αναζητήσουμε είναι το να υπάρξει ισοδυναμία. Ε, το να επιβάλλουμε την ισοδυναμία σε όλους τους τομείς δεν φαίνεται να είναι κάτι αναγκαίο. Βεβαίως έχουμε τη δέσμευση των G20 ιδιαίτερα για τα παράγωγα, κάτι που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και ε, κυρίως ε, λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια που έγιναν από τον Επίτροπο όταν μίλησε στο ε, Ινστιτούτο Διεθνών Τραπεζιτών. Θα πρέπει να έχουμε τη βεβαιότητα ότι υπάρχει αναγνώριση συγκρίσιμης ε, νομοθεσίας. Θα ήθελα να ζητήσω από τους σχεδόντες ε, εισηγητές να υποστηρίξουν τις τροπολογίες αυτές που αφορούν τις μεταβατικές ρυθμίσεις και που δίνουν προτεραιότητα σε ορισμένες χώρες έτσι ώστε να υπάρχει ε, εποπτεία της αγοράς. Περιορίζω τα σχόλιά μου σε αυτό νομίζω ότι ο εισηγητής προχώρησε πάρα πολύ το θέμα αυτό και έγινε ένας ιδιαίτερα επικοδομητικός διάλογος. Είναι εντυπωσιακό το, τη συμφωνία που επετεύθη. Είναι δυνατόν να ακολουθήσουμε το χρονοδιάγραμμα λαμβάνοντας υπόψη το σημείο στο οποίο έχουμε φτάσει. Πιστεύω ότι οι τομείς διαφοράς θα καταφέρουν ε, δεν θα, ε, δεν μπορέσουν να γεφυρωθούν. Μερικές φορές είναι θέμα ιδεολογικών διαφορών. Λαμβάνοντας υπόψη τον θέμα των παραγωγών, συμφωνώ με το στόχο του εισηγητή ε, να γίνει κατά τη διάρκεια των διακοπών του καλοκαιριού. Πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε και ενδεχομένως στο τέλος θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ πολύ. Γιόγκεν από τον Ευχαριστώ. Καταρχάς, ε, να ευχαριστήσω τον ε, Μάρκους Φέμπερ. Θεωρώ ότι δούλεψε με ανοιχτό και δίκαιο τρόπο και σε επίπεδο περιεχομένου θεωρώ ότι υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία και για μας συζητούνται γιατί ε, πάντοτε υπάρχει μια πίεση ως προς αυτά τα θέματα. Καταρχάς να πω κάτι για τα άτομα που ήταν εδώ για τι μη κυβερνητικέ οργανώσει. να ε, υπογραμμίσω αυτό που είπαν και προηγούμενοι. Αυτό το θέμα είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα στην ε, Γερμανία τα τελευταία χρόνια σχετικά με την ε, κερδοσκοπία ως προς τα τρόφιμα. Υπάρχει θέμα υπαρξιακό. Κανείς αν ε, δεν μπορεί να φάει, στην ουσία δεν μπορεί να επιβιώσει. Είναι ένα θεμελιώδες ε, θέμα, ε, το θέμα της ε, δυνατότητας πληρωμής των τροφίμων και πραγματικά είναι ένα δραματικό ζήτημα το οποίο μέσα στα πλαίσια της Ευρώπης, της ποιότητας ζωής που έχουμε εδώ και της του πόσο ακριβά είναι κάποια ζητήματα, ε, κάποια προϊόντα. Μας ε, αγγίζει ιδιαίτερα. Είναι η Εκκλησία η οποία εμπλέκεται σε αυτό το θέμα και στο μεταξύ ο καθένας εκφράζει ε, πολλές απόψεις για αυτό το θέμα. Να υποστηρίξω λοιπόν αυτό που υπόθηκε ότι είναι μια πολύ σοβαρή ιστορία και υπάρχει ένα κομμάτι της, του κοινού που ενδιαφέρεται πάρα πολύ για, για αυτά που συμβαίνουν εδώ. Είναι ε, πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό το ζήτημα και αν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν ε, ε, ιδέες για τη βελτίωση του κόσμου, όπως είπε και ο Μάρκος Φέμπερ, είναι καλό να τις υποστηρίζουμε και να τις συζητούμε τουλάχιστον. Θεωρώ ότι αυτό που γίνεται με αυτές τις διαμαρτυρίες δεν είναι χειρότερο από αυτό που κάνουν κάποια λόμπι. Και επίσης αυτό με τα email που είπατε θεωρώ ότι είναι λίγο ε, καταπιεστικό αλλά στη δημοκρατία πρέπει επικοδομητικά να λύνουμε τέτοια ε, προβλήματα. Ε, δεν είναι προσωπική επίθεσή μου, είναι απλώς η δική μου συμβουλή σε ένα σημαντικό ζήτημα. Να πω τώρα για τα όρια θέσεων. Έχουμε συγκεκριμένες αυστηρούς κανόνες και συγκεκριμένες αυστηρές προτάσεις να πω ότι δεν έχει να κάνει με συγκεκριμένες ε, μεθόδους που πρέπει να διατηρηθούν. Έχουμε κάποιους ε, στόχους για μείωση της κερδοσκοπίας, καλύτερη ρύθμιση. Εκεί είμαστε ανοιχτοί. Είναι μέσα στο νόημα της συζήτησή μας ε, να συνεννοηθούμε σχετικά με το ποιες είναι οι μέθοδοι που θα είναι οι κατάλληλες για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς να πω ότι η κερδοσκοπία ε, δεν πρέπει να, ε, θα πρέπει να περιοριστεί και να ελεγχθεί. Άρα δεν υπάρχει βασική διαφωνία. Το θέμα είναι μόνο οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν. Για τη διαφάνεια, ναι. Και αυτή τη θεωρούμε σημαντική. Για μας ε, είναι σημαντικό τα δεδομένα των συναλλαγών θα πρέπει τακτικά να δημοσιεύονται για το θέμα της προστασίας των καταναλωτών. Για μας ε, είναι σημαντικό να μην υπάρχουν μόνο ε, συγκεκριμένες, ε, συγκεκριμένοι περιορισμοί για τα κίνητρα, αλλά θέλουμε να υπάρχει ένας ξεκάθαρος ε, ορισμός ε, της ανεξάρτητης παροχής συμβουλών και να υπάρχουν ε, εναλλακτικές ως προς την παροχή κινήτρων σε επίπεδο Ευρώπης. Ο στόχος πρέπει να είναι ένα μοντέλο λογικό. Για την απαγόρευση συμφωνώ με αυτό που είπε ο Μάρκος Φέμπερ. Το συζητήσαμε ήδη ε, κατηδίαν. Όταν εκ των πρωτένων δίνεται άδεια, ε, νομιμοποιούνται κάποια πράγματα και αυτό ε, δεν πρέπει να γίνεται. Δεν ξέρω αν γίνεται κανείς ε, να πάρει πίσω αυτό που έχει ήδη επιτρέψει. Άρα θα πρέπει λίγο πολύ να δούμε πώς θα επέμβουμε ώστε να μην πάμε προς την ε, λάθος κατεύθυνση. Αυτές οι άδειες λοιπόν είναι ένα νέο πρόβλημα. Το τέλος θέμα, το τελευταίο θέμα είναι ε, τα, οι μηχανισμοί υψηλής συχνότητας ποιο είναι το νόημά τους. Ε, τεχνικά είναι δυνατό, αλλά ό,τι είναι τεχνικά δυνατό έχει και νόημα. Ε, δεν μπορούμε να ε, απαλλαγούμε από τον υπολογιστή, όπως είπε και ο Φέμπερ, όμως ε, όλες αυτές οι συναλλαγές με το κομπιούτερ ε, γίνονται δύσκολες. Εδώ να πω, όπως και ε, υπογράμμισαν και οι άλλοι ότι πρέπει να, μειωθεί αυτή, να μειωθούν αυτές οι συναλλαγές υψηλής συχνότητας. Ε, ο, ο τρόπος που προτείνει ο συγγιστής ε, με την μεγαλύτερη διάρκεια είναι κάτι που μπορεί να συζητήσουμε αν είναι σωστό. Ο στόχος είναι να μην γίνεται κατάχρηση σε αυτόν τον τομέα γενικά να περιοριστεί στο μίνιμουμ γιατί χωρίς να αυξηθεί ο χρόνος ε, με αυτές τις υψηλές συχνότητες συναλλαγές έχει δεκαπλασιαστεί ο τζίρος. Είναι ένα θέμα λοιπόν πολύ ε, δύσκολο και να πω ότι πρέπει να κατανοήσουμε τους πολιτικούς στόχους μας και να συζητήσουμε ποιες είναι οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιήσουμε για αυτούς τους στόχους. Στις συζητήσεις ως τώρα ε, που έχουν γίνει για τα θέματα της υψηλής συχνότητας, αυτό είναι πάντοτε το ζήτημα. Αυτά ήταν οι παρατηρήσεις μας. Οι παρατηρήσεις μου ευχαριστώ πολύ. Okay, thank you very much. Σας ευχαριστώ. Έχω ακόμη έξι συναδέλφους που θέλουν το λόγο. Για να δούμε αν θέλει κάποιος άλλο το λόγο. Πείτε Σίμον Μπέρκαλμπερκ. Εγώ είμαι η τελευταία που ζήτησα το λόγο. Θέλει κανείς άλλος να λάβει το λόγο. Εάν όχι, έχει καλώς. Αρχίζουμε με τον Πίτερ πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την ε, εμπεριστατωμένη παρουσίαση που έκανε και θα ήθελα να αναφέρω ένα θέμα που και εκείνο ανέφερε. Και θα επικεντρωθώ σε αυτό δεδομένου ότι έχουμε καθυστερήσει μετά από αυτά τα οποία είπαν ο Ίγκο και Κλούτ. Η ανεξαρτησία των, ε, των οικονομικών συμβούλων είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό, αλλά δεν τηρείται συχνά. Εκεί που λέει η Κομισιό ε, ανεξαρτησία του Συμβούλου, θα πρέπει όντως να το θέσουμε σε εφαρμογή. Δεν θέλω να δημιουργήσω προβλήματα, αλλά δεν... Νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε τον σαφή ορισμό αυτού του Οικονομικού Συμβούλου για να ξέρουμε όχι πώς θα τον ε, ανταμείψουμε, αλλά τι ακριβώς πρέπει να κάνει. Τροπολογία 735. Εκεί λέει ότι ε, έχουμε να κάνουμε με ανεξάρτητο σύμβουλο και θα ήθελα να μας πει η Κομισιόν πώς ακριβώς το εννοεί. Για να υπάρχει πραγματική ανεξαρτησία θα πρέπει οποιαδήποτε η ηλική ή άλλου τύπου ανταμοιβή να απαγορεύεται για να είναι πραγματικά ο σύμβουλος ανεξάρτητος. Ο ορισμός λοιπόν αυτός θα πρέπει να δοθεί με σαφήνεια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είπαμε ότι υπάρχει στην ε, τροπολογία 747. Επαναλαμβάνω, θα πρέπει να είναι σαφής ο ορισμός αυτού του Συμβούλου, ώστε να μπορεί να είναι προστατευμένος ο κάθε πελάτης, ο κάθε καταναλωτής. Ευχαριστώ. Ο Μπούρκαρτ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την εξαιρετική εργασία του. Και εγώ είχα την τύχη, μεταξύ άλλων, να έρθει στην εκλογική μου περιφέρεια, το Στρασβούργο, μία ομάδα δημοσιογράφων και μου ζήτησε διάφορες πληροφορίες για αυτά τα θέματα. Κάποιοι κανόνες όμως γίνονται στο κοινοβούλιο και όχι από τους δημοσιογράφους. Γι' αυτό και εγώ ως ε, ευρωβουλευτής θα λέω την άποψή μου ελεύθερα. Θέλω να αναφερθώ σε αυτά τα θέματα της ε, αμοιβή των συμβούλων σε θέματα Η προσέγγιση του Μάρκους θα μας επιτρέψει να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια, πράγμα που θα βοηθήσει στην επιλογή του τον πελάτη. Σήμερα όμως πρέπει να σας πω ότι η μικρή Επενδυτέ δεν γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τους κανόνε και τι διατάξει. Γι' αυτό νομίζω θα πρέπει να τους βοηθήσουμε. Η προσέγγιση του εισηγητού λοιπόν πιστεύω ότι πάει στη σωστή κατεύθυνση. Η προμήθεια και η αμοιβή του Συμβούλου θα πρέπει κατά την άποψή μου να επιτρέπονται. θα πρέπει να ακολουθήσουμε ένα ρεαλιστικό πρότυπο, γιατί αν περάσουμε από ενός τύπου συστήμα ε, από τη μια στην άλλη, δεν θα κατορθώσουμε τίποτα. Θα πρέπει να προβλέψουμε μία μακρά μεταβατική περίοδο και αν ε, ασχοληθεί κανείς με τα διάφορα επενδυτικά προϊόντα στην αγορά, θα συνειδητοποιήσει ότι δεν υπάρχει μεγάλη σαφήνεια μεταξύ των προϊόντων αυτών, ώστε να επιτρέπεται να δοθεί κάποια συμβουλή έναντι αμοιβή. Ένας καταναλωτής που θα πρέπει να ε, προστρέξει σε ένα σύμβουλο πληρώνει δύο φορές την αμοιβή του και την ε, ε, προμήθειά του. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να συστήσουμε ένα παράλληλο σύστημα. Δηλαδή και ο πελάτης και ο ενδιάμεσος, ο διαμεσολαβητής, συγγνώμη, θα πρέπει να αποφασίσουν μεταξύ τους πώς θα διαμορφωθεί η αμοιβή. Διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα αυτό. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία νομίζω ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να αποσαφινιστούν και συμφωνώ και με κάποιους από τους προλαλήσαντες που είπαν ότι το θέμα της διαμόρφωσης των τιμών των πρώτων υλών και των ειδών διατροφής είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να χειριστεί ο συνάδελφος με μεγάλη δεξιοτεχνία και ακρίβεια στην εκθεσή του. Γιατί θα πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο θέλουμε να προχωρήσουμε. Διότι για πολλά άτομα η ποιότητα της ζωής, η επιβίωσή τους εξαρτάται από αυτά τα θέματα. Γι' αυτό συμφωνώ με αυτά που πάνε προηγουμένως οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ. Η κυρία Λούλινγκ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ως ε, Κοσμήτερος θα ήθελα μετά από αυτό που είπε ο κ. Σνούτε να πω τα εξή. Για αυτό το οποίο συνέβη προηγουμένως. Κανένας ε, δεν μπορεί να κάνει τέτοιου είδους ε, ε, επεισοδιακές εισόδους στην Ολομέλεια. Υπάρχουν κανόνες με τους οποίους μπορεί κανείς αν θέλει να διαμαρτυρηθεί. Και υπάρχουν κανόνες ασφαλείας. Εδώ όμως θα πρέπει να κάνουμε κάτι για να δούμε πώς η μικρές αίθουσες στις οποίες συνεδριάζουμε μπορούν να προστατευτούν από τέτοιου είδους ε, γεγονότα. Για να μπορέσουμε λοιπόν να είμαστε σίγουροι για την δική μας ασφάλεια. Δεν θα πρέπει να επιτρέπουμε τέτοιου είδους επεισοδιακές εισόδους σε αίθουσες, γιατί μπορεί να γίνουν και χειρότερα πράγματα. Παρακαλώ. Έχω μία ερώτηση για την κυρία Λούλινγκ. Όντως, εάν θέλετε, μπορούμε να πούμε ότι ευτυχώς δεν υπήρξε ε, βία, διότι αν υπήρχε τέτοιου είδους φαινόμενο, ε, θα ήταν σοβαρά τα πράγματα. Εγώ δεν αισθάνθηκα όμως απειλή καμία στιγμή. Βεβαίως δεν σεβάστηκαν τους κανόνες, είναι αλήθεια. Αλλά δεν υπήρξε πράξη βίας. Η βία τι είναι. Να υπάρχει και στα είδη διατροφής και κάποιος να μην μπορεί να φάει και να πεθάνει. Εδώ δεν είδαμε καμία βία να ε, βία το ότι αντιστάθηκαν στους κλητήρες δεν τους είδατε ίσως, λέει η κυρία Λούλη. Και αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν την αίθουσα. Εγώ τους είδα όμως. Είδα ότι οι κλητήρες χρειάστηκε να τους σπρώξουν για να τους βγάλουν από την αίθουσα. Δεν το δα, δεν το δα. Εν πάση περιπτώσει, ακούστε, λέει η πρόεδρος, Είπα ότι πρέπει να σέβονται τους κανόνες, λέει η κυρία Λόλιν. Διότι το προσωπικό του Κοινοβουλίου υπέστη, πράξη, υπέστη βίας εκ μέρους τους όταν αρνήθηκαν να, κάνουν, ε, να βγουν από την ασφάλεια. Ακούστε, δεν κάνουμε συζήτηση εδώ για την βία και για το πώς μπήκαν και πώς βγήκαν. Ε, μιλάμε για το θέμα που μας απασχολεί και έχουμε και πολλή συζήτηση. Όταν τελειώσει η συζήτηση για τον κανονισμό ΜΥΦΙΤ, μπορούμε αν θέλετε και έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε. Λίγη συζήτηση για αυτό το θέμα. Πιστεύω ότι είναι λυπηρό το ότι υπήρχε τέτοιου είδου ε, λόμπι επιθετικό και υπήρχαν και προσπάθειες ε, ε συνεργασμού για κάποιους από εμάς. Σε πάση περιπτώσει, ας επανέλθουμε άστριτ στο θέμα μας και συνεχίσουμε, λέει η Πρόεδρος. Παρέμβαση της κυρίας Λούλιν χωρίς μικρόφωνο. Ναι, δεν έκανα εγώ τη συζήτηση. Άλλοι να, ο άλλος ήθελε να απαντήσει για τους κανόνες. Τέλος πάντων. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ τον Μάρκους Φέρμπερ για τη δουλειά που έκανε. Εγώ πολύ σύντομα θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια θέματα. Πρώτα απ' όλα στο θέμα της πολυπλοκότητας των προϊόντων. Είναι κάτι το οποίο οδήγησε ορισμένους συναδέλφους στο να καταθέσουν ε, τροπολογίες. Για την διανομή τώρα των προϊόντων, η έννοια του κινδύνου δεν έχει απαραίτητα σχέση με την πολυπλοκότητα. Κυρίως για την ε, χρησιμοποίηση των παραγόγων προϊόντων που είναι λιγότερο επικίνδυνα. Υπάρχουν άλλα προϊόντα τα οποία οι ιδιώτες επενδυτές έχουν ενημερωτικά έγγραφα σύντομα και ενημερωτικά ώστε να μπορέσουν να καταλάβουν σε ποιο προϊόν επενδύουν. Άρα δεν νομίζω ότι πάντα πρέπει να το συνδέουμε το θέμα με την πολυπλοκότητα. Τώρα, το θέμα του inducement και των αμοιβών. Θα ήθελα εγώ να συγχαρώ τον ε, ε, εισηγητή ο οποίος θέλει με διαφάνεια να γίνονται τα πάντα ώστε να διευκολυνθούν, να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην ενημέρωση. Ε, αυτό νομίζω ότι είναι η καλύτερη λύση. Διαφορετικά, ε, οι μικροϊδιώτες επενδυτές θα απομακρυνθούν από τις αγορές. Μάρκος Φέμπρε ξέρει πώς ε, λειτουργούν οι αγορές και η συστηματικοί εσωτερικοποιητές θα πρέπει να ξέρουν τι κάνουν και να παρέχουν το καλύτερο και το πλέον κατάλληλο και πιο διαφανές σύστημα. Νομίζω επίσης ότι για τα μη ε, μετοχικά ε, προϊόντα θα πρέπει η να υπάρχει διαφάνεια και στις προσυναλλακτικές συναλλαγές. Επίσης, το θέμα αυτό του τόπου διαπραγμάτευσης σε κεντρικούς αντισυμβαλόμενους θα πρέπει ε, να οριστεί ώστε να μην υπάρχουν πρόσβαση πολλών στην ίδια πλατφόρμα, στον ίδιο τόπο, ώστε να αυξάνεται το ρίσκο. Αυτά ήθελα να πω και να ευχαριστήσω τον Μάρκος ακόμη μια φορά για την προσέγγιση του και για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τις διάφορες τροπολογίες. Υπάρχουν πάμπολες, αλλά νομίζω ότι θα κατορθώσει να μας οδηγήσει σε πολύ καλές συμβαστικές τροπολογίες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, ο Γουλφ. Ευχαριστώ να πω σύντομα ότι ε, αυτή η οδηγία ε, είναι πολύ σημαντική και ότι πραγματικά θα θέσει τους κανόνες παιχνιδιού στο μέλλον. Αλλά αυτό δεν είναι εγγυημένο. Βλέπετε στην Ευρωζώνη πώς γίνονται τα πράγματα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ολοκλήρωση και ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι ο Κάμερον τον Δεκέμβριο ήδη είχε αναφέρει το θέμα ε, των χρηματιστηρίων στο Λονδίνο, άρα δεν υπάρχει καμία ε, ε, εγγύηση ότι θα πάμε στο μέλλον προς μία κατεύθυνση και όχι σε πολλές. Άρα για μας αυτή η οδηγία έχει πολύ μεγάλη σημασία. Κάποια βασικά σημεία για τις ε, βιομηχανικές επιχειρήσεις νομίζω ότι έχω άλλη άποψη από τον εισηγητή. Αυτό είναι θέμα της Ήτρε. Ε, αυτό που είπατε για ε, ένα θηγατρικό προϊόν των βασικών αγαθών, ας πούμε, που θα πρέπει να το εξετάσουμε, να δούμε ποιες είναι οι ε, οι δράσεις του ε, ε, στην πραγματική οικονομία. Να πω επίσης ότι γενικά αυτό που είπε ο συνάλφος Μπάλς αλλά και ο εισηγητής σχετικά με, τις, με τα κίνητρα της προμήθειας βλέπουμε ότι στην πράξη οι τράπεζες έχουν ένα πολύ ωραίο τρόπο αυτή τη στιγμή να συσσωρεύουν προμήθειες για τα δικά τους προϊόντα όπως τα λένε και πάντοτε είναι κατά ε, ανταγωνιστικών προϊόντων ε, που πολλές φορές ε, θα ήταν προς συμφέρον του πελάτη. Έτσι λοιπόν, όσον αφορά τις διάφορες κατηγορίες προϊόντων, νομίζω, ας πούμε για το usage, ότι πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ της complex και non-complex, πολύπλοκης και μη πολύπλοκης χρήσης. Αυτό θα πρέπει να είναι στα προϊόντα και όχι εδώ. Ε, πρέπει να το συζητήσουμε για να βρούμε λύση. Όσον αφορά στις τρίτες χώρες, ε, εγώ ως ε, μέλος του Άλντε, αντίθετα με τον συνάδελφό μου, που είναι υπέρ μιας φιλελεύθερης πρόσβασης, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει εναρμονισμός των ευρωπαϊκών μεν να υπάρχει περιορισμός της ευρωπαϊκής παρεμβολής, αλλά να μην ε, απαγορεύονται συναλλαγές, να είναι ο πελάτης ε, που θα έχει την πρωτοβουλία. Το, οι συναλλαγές υψηλής συχνότητας είναι κάτι τόσο τεχνικό που πραγματικά δεν ξέρω ε, τι γίνεται στην πράξη. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των 5 και των 500 εκατοστών του, χιλιο, του δευτερολέπτου δεν ξέρω αν μπορούμε πραγματικά να έχουμε μια λογική θέση για αυτό το θέμα, για, τα, ε, για τις προμήθειες, για αυτά που είπανε, για τα τέλη μάλλον που έθεσαν το θέμα οι συνάδελφοι, ότι θα ήθελα να πω ότι καλό θα ήταν ε, ναι με να υπάρχει μία συζήτηση με τους ειδικού, αλλά από την πλευρά μας θα πρέπει εμείς να πάρουμε αντικειμενικές ε, πληροφορίες ε, από τους ειδικού. Νομίζω ότι ο κόσμος δεν ξέρει ότι το 97% όλων αυτών των ε, συναλλαγών γίνεται στο Σικάγο και μόνο το υπόλοιπο στην Ευρώπη. Άρα θα πρέπει να βρούμε σωστές εξειδικευμένες πληροφορίες από αυτούς που είναι ειδικοί. Τώρα για αυτό που είπε ο εισηγητής για τις πράξεις κατά εξουσιοδότηση, δεν είναι το μόνο θέμα στην Ευρώπη που προσπαθούν να ε, χρησιμοποιήσουν με λάθος τρόπο ε, το θέμα των πράξεων κατά εξουσιοδότηση. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αρλίν. Θα είμαι σύντομη. Γιατί ήδη μίλησε εξ ονόματος της ομάδας. Απλά και μόνο θα ήθελα να τονίσω το θέμα της προστασίας του επενδυτή. Μολονότι γιατί άκουσα σαφώ από τον εισηγητή ότι δεν θέλουμε κατά ανάγκη να ακολουθήσουμε το παράδειγμα μια συγκεκριμένη χώρα μέλο. Θα πρέπει όμω να έχουμε κατά νου τις καταστροφές που επήλθαν σε ορισμένε χώρε μέλη σαν αποτέλεσμα τη νήσης προστασία των επενδυτών. Στι τροπολογίε μου λοιπόν εστιάζομαι στο θέμα τη αποκάλυψης πληροφοριών, τη κοινοποίηση πληροφοριών υπέβαλα τροπολογίες για την ανάγκη περαιτέρω προστασίας των καταναλωτών και των επενδυτών διασφαλίζοντας ότι οι εταιρείε επενδύσεων δεν θα έχουν μια συμπεριφορά η οποία να μην είναι προς το καλύτερο συμφέρον των πελατών τους ή να βοηθούν, να ευνοούν ένα συγκεκριμένο χρηματοδοτικό μέσο σε περίπτωση που ένα άλλο ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του πελάτη. Ο πελάτης θα πρέπει να έχει τις καλύτερες δυνατές πληροφορίες, το κόστος της συμβουλευτικής, το τίμημα, την τιμή που θα πρέπει να καταβάλει δεν θα πρέπει να δέχονται προμήθειες ή να έχουν απολευές από ένα τρίτο μέρος ή από κάποιον που δρά εξ ονόματος κάποιου άλλου. Θα πρέπει να πληρώνονται εξ ονόματος του πελάτη. Νομίζω ότι υπάρχει σαφής ανάγκη να δηλωθούν στον πελάτη τα απαιτούμενα ποσά. Τα ποσά αυτά ε, να παρουσιάζονται ξεχωριστά από άλλα οφειλόμενα ποσά θα πρέπει να ενημερώνει το πελάτη όταν υπάρχει κάποια άλλη εταιρεία η οποία καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες ε, του πελάτη Πιστεύω ότι αυτά είναι βασικά προαπαιτούμενα που αφορούν την ενημέρωση για την αποκάλυψη πληροφοριών και ελπίζω ότι ο εισηγητής θα μπορέσει να τα εντάξει στον τελικό συμβιβασμό. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι η ώρα μας πιέζει. Θα ήθελα όμως να μιλήσω για αυτό το θέμα και εγώ. Πιστεύω ότι ο εισηγητής, όπως είπαν όλοι, ε, έκανε μια εξαίρετη δουλειά. Πραγματικά θα πρέπει να κάνουμε κάτι που θα σταθεροποιήσει τις αγορές. Ένα θέμα που θα ήθελα να αναφέρω αφορά την αγορά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δεν θα πρέπει να την περιορίσουμε ιδιαίτερα αυτή την αγορά και ενδεχομένω θα ήταν κρίσιμο για τον εισηγητή να έχει κάποια συζήτηση σχετικά με τα όσα γίνεται ε, ε, κάνουμε με το venture capital. Θα πρέπει να γνωρίσουμε ότι αυτό θα μπορούσε να αναπτυχθεί και ότι υπάρχει ανάγκη να κάνουμε κάτι. Συμφωνώ με αυτό που είπε και, σχετικά, και είμαι σχετικά με αυτό το θέμα. Θα πρέπει να έχουμε τη βεβαιότητα ότι μεγιστοποιούμε τις ευκαιρίες ανάπτυξης. Μερικές φορές αναπτύσσεται κανείς ως ένα σημείο και ε, χρειάζεται περισσότερη ε, νομοθεσία. Ας συνεχίσουμε λοιπόν να κάνουμε αυτά που κάνουμε με το ε, venture capital, με το επιχειρηματικό κεφάλαιο. Επίσης αναφερθήκαμε στα λανθασμένα κίνητρα. Είπαμε, αναφερθήκαμε στους επενδυτές, ε, αναφερθήκαμε σε κρυφές αμοιβέ διαχείρισης. Ο επενδυτής μπορεί να επιλέξει μία λανθασμένη επένδυση γιατί πιστεύει ότι του αποφέρει περισσότερα και να την προτιμήσει αντί για μία μακροπρόθεσμη επένδυση. Συμφωνώ με όσα είπατε ως προς τα μέτρα που λαμβάνονται στην οδηγία περί κεφαλαίων. Θα μπορούσαμε να ανακυκλώσουμε μερικές από τις τροπολογίες που ήδη υπάρχουν στο κείμενο του Κοινοβουλίου που αναφέρεται στα ρέπος και συμφωνώ με την άποψη του εισηγητή ότι θα μπορούσαμε να αντιγράψουμε όσα έχουν συμπεριληφθεί σε άλλες οδηγίες και, έχουν αποδειχθεί, και έχει αποδειχθεί ότι ήταν ορθά. Τώρα σε ό,τι αφορά το, το θέμα των επενδύσεων, μιλώντας για μια καλύτερη αντιμετώπιση των επενδυτών, πολλές φορές καταλήγουμε σε ένα κατακαιρματισμό και σε μια διαδικασία εξυγίασης. Αυτό όμως θα πρέπει να το καθοδηγεί η αγορά. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να διατηρήσουμε την ισορροπία που έχει επιτευχθεί και η οποία δεν καταλήγει όμως σε διαλειτουργικότητα. Νομίζω ότι θα πρέπει να ζήσουμε και ε, να αφήσουμε και τους άλλου να ζήσουν. Υπάρχει εν γενός η δυνατότητα αναζήτησης παρέμβασης εάν υπάρχει κίνδυνος αποσταθεροποίησης και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το κατά πόσον θέλουμε μία ρυθισμισμένη αγορά ή αν θέλουμε συστημικούς κινδύνους. Στο παρελθόν θεωρούσαμε ότι ε, τα big banks ήταν μια καλή ιδέα. Αλλά τώρα νομίζω ότι θα πρέπει να πάρουμε σοβαρά το θέμα του ανταγωνισμού και της ανταγωνιστικότητας. Θα έλεγα ότι εδώ δίνεται ένας υπαρξιακός αγώνας για το ευρώ και θέλουμε η Ευρώπη να είναι αξιόπιστη. Θα πρέπει λοιπόν να μιλάμε για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα αλλά και να εφαρμόζουμε τα όσα λέμε. Θα πρέπει να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι στη συνθήκη άρθρο 119 αναφέρεται ρητός ότι οι οικονομικές μας πολιτικές θα πρέπει να προωθούνται με βάση τις αρχές της ελεύθερης αγοράς και της αγοράς του ελεύθερου ανταγωνισμού. Αυτό αναφέρεται στο άρθρο 119, να σας θυμίσω. Παρόλο το ευρώ, θα πρέπει να διατηρηθεί ως στόχο να διατηρηθούν οι γενικέ πολιτικέ στην Ευρώπη σύμφωνα με τι αρχέ τη οικονομία ελεύθερη αγορά σε πλαίσια ελεύθερου ανταγωνισμού. Νομίζω ε, ότι δεν χρειάζεται κανένα opt-out δεν αρχίσουν να, τεθούν, να τίθεται θέματα με το ευρώ. Όταν κοιτάξουμε το θέμα τη ε, διακυβέρνηση, θα πρέπει να πούμε ότι έχουν εισαχθεί ήδη μεταρρυθμίσει σε διάφορους τομεί. Επτά χώρε ε, κάνουν μια σαφή αναφορά σε αυτό στι τάσει. Η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Κύπρο, η Φιλανδία και η Αυστρία. Όλε ε, ξέρουν ότι θα πρέπει να καταφέρουν περισσότερα στον το μέα των υπηρεσιών. Βεβαίω, δεν θέλω να κάνω κανένα παραλληλισμό. Σας παρακαλώ λοιπόν ας ε, ας κάνουμε μια προσπάθεια να βάλουμε μαζί την ομοθεσία, τις συνθήκες, την, την ε, διακυβέρνηση. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, θέλουμε να αναπτυχθεί η Ευρώπη και σε αυτή τη βασική νομοθεσία θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ακολουθήσουμε αυτές τις αρχές και να τις υποστηρίξουμε. Διαφορετικά κανένας δεν θα μας πιστέψει, οι αγορές δεν θα μας πιστέψουν και βεβαίως μπορεί να κατσουφιάσουν και οι G20. Ευχαριστώ και λόγω στον Μάρκος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, να πω ε, καταρχάς ότι ευχαριστώ τους συναδέλφους και ελπίζω ότι ε, αυτή η θετική ας πούμε στάση που επέδειξαν σε όλες τις παρεμβάσεις τους θα μας βοηθήσει στην εργασία μας. Να κάνω κάποιες σύντομες παρατηρήσεις και το θέμα έκλεισε για μένα. Και εγώ... Τις τελευταίες εβδομάδες ε, συζήτησα με πολλούς ε, ε, στο γραφείο μου. Έγινε ανταλλαγή επιχειρημάτων και δεν είναι καλύτερο το επιχείρημα όταν επιλέγεται άλλη μορφή παρουσίασής του. Νομίζω λοιπόν ότι είναι καλό καθένας από ε, να δέχεται έναν συνομιλητή και να κατατίθενται επιχειρήματα ε, τα οποία ε, δεν είναι απαραίτητο ε, χειρότερα από ότι μια τράση διαμαρτυρίας εδώ. Αυτό λοιπόν που βλέπω είναι ότι η παρουσίαση δεν παίζει κανένα ρόλο, το αντίθετο μάλιστα. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα που πρέπει να απαντήσουμε. Ε, συζητήσαμε το θέμα των ε, οργανισμένων μηχανισμών διαπραγμάτευσης. Το είπαν πολλοί συνάδελφοι και έκαναν προτάσεις ε, σχετικά με έναν συμβιβασμό που θα μπορέσουμε να πετύχουμε. Θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα όσον αφορά τι συναλλαγέ υψηλή ε, συχνότητα, ε, ξέχασα στην παρουσίασή μου να αναφέρω το θέμα της απογόρευσης της sponsor taxes. Ε, είναι ένα συγκεκριμένο θέμα που έχει να κάνει με μια διαφανή και χωρίς ρυθμίσεις πρόσβαση έτσι ώστε να υπάρχουν οι τεχνικές προϋοθέσεις ώστε οι συναλλαγές να γίνονται σε μια τέτοια κατεύθυνση Παρακαλώ ε, να μην μιλάτε τόσο δυνατά, Άστριντ. να πηγαίνουν οι συναλλαγές ε, σε τέτοια κατεύθυνση ώστε τελικά ε, να μην είναι προς το συμφέρον των συναλλασσόμενων. Όσον αφορά στις εξαιρεσει, το είπατε κι εσείς, Ξεκινάει και πάλι αυτό το θέμα για μένα ε, φαίνεται ότι ναι μεν πρέπει να υπάρχουν ε, εξαιρέσεις αλλά αυτό που έχει επιλέξει η Κομισιόν ε, ως ορισμό για το κεφάλαιο είναι πραγματικά αυτό που θα ανοίξει τον ασκό του αιώλου. Πρέπει να το συζητήσουμε γιατί η κάθε τράπεζα θα μπορεί να πει ότι θα εμπλακεί σε αυτό το σύστημα και έχω πραγματικό ενδιαφέρον. Το λέω λίγο σκληρά, είναι λίγο πολύπλοκο. Αλλά ε, ε, αν, ε, αν ο καθένας στην Γερμανία θεωρεί ότι μπορεί να ανοίξει έναν τόπο διαπράγμα, επειδή δεν υπάρχει ε, ρύθμιση ε, τότε και δεν υπάρχει και ανταγωνισμός, τότε ε, κρατικά, σε επίπεδο κρατικό, τότε ε, θα προκύψουν μονοπόλια. Και αυτό είναι ενάντια στο συμφέρον των πελατών. Πρέπει λοιπόν να λύσουμε αυτό το ζήτημα. Εν είμαστε στο κρατήδι Άμμο, ας πούμε, στην πρωτεύουσα που υπάρχει ένας ε, πολιτικός σχηματισμός ε, που θέλει να χρησιμοποιήσει αυτά τα εργαλεία ε, δηλαδή να υπάρχει προστατευμένη εργασία και να υπάρχει μονοπόλιο και μετά καταλαβαίνετε ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει γιατί το επιχειρηματικό μοντέλο ενός κρατικού οργανισμού δεν ταιριάζει με κάτι τέτοιο. Άρα ε, πραγματικά να ρωτιέμαι αν είναι αυτό η σωστή προσέγγιση. Και έχω αμφιβολίες αν είναι ε, σωστό τώρα για την ε, complex paper usage, την πολύπλοκη χρήση εγγράφων. Δεν θεωρώ ότι η χρήση, το usage είναι η λύση του προβλήματος αν είχαμε τα πάντα τυποποιημένα στο usage, θα βλέπατε ότι τελικά ήταν τα είναι τα προϊόντα που ε, είναι σημαντικά για τους κανονικούς ε, τους ε, επενδυτές. Υπάρχουν πάντοτε προϊόντα που ταιριάζουν στους μικρούς επενδυτές. Και το usage είναι απλώς μια προσπάθεια να έχουμε ε, τυποποίηση. Το use το έχουμε συζητήσει πολλές φορές ε, ότι χρειαζόμαστε διαφάνεια. Με το usage ε, τώρα να λυθούν τα προβλήματα είναι λάθος. γιατί είναι πολύ πέρα από αυτό που εμείς θεωρούμε ως ε, ε, σωστή προστασία των καταναλωτών. Κατά τα άλλα, χαίρομαι για τα όσα υπόθεσαν από τους, υπόθηκαν από τους άλλους, ε, από τους κοιόδης. Τα συζητήσαμε και τις ομάδες. Ε, νομίζω ότι μπορούμε επικοδομητικά να συνεχίσουμε και γι' αυτό ευχαριστώ ε, για τις πολλές παρεμβάσεις, όχι τόσο για τις τροπολογίες όσο για τις ε, παρεμβάσεις σας, το ότι πήρατε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Είχα τη φιλοδοξία να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα, αλλά ο χρόνος μας πιέζει. Για να δούμε. Λέμε να ψηφίσουμε στην Επιτροπή στις 9 ή 10 Ιουλίου και δυνητικά το Σεπτέμβριο, εάν ο Μάρκος θα μπορούσε να διατηρήσει την ταχύτητα, την εντυπωσιακή ταχύτητα που έχει αναπτύξει. Περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα της ημερησίας ε, διάταξης που αφορά τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς. Η Αλήν Μακάθρη είναι η εισηγήτρια και για τα δύο αυτά θέματα. Θα ήθελα να κάνω μία ανατείνωση, μόνο ότι είναι για το δεύτερο θέμα, ότι έχουμε συμφωνήσει με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για την οδηγία και κατά συνέπεια θα δοθεί και πάλι η δυνατότητα κατάθεσης τροπολογιών και από αυτή την Επιτροπή. Η προθεσμία έκλεισε πριν επιτευχθεί αυτή η συμφωνία. Η Ερλίν όμως έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συναδέλφους που μπήκαν ε, στον κόπο να ασχοληθούν με το τόσο πολύπλοκο αυτό θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις τροπολογίες που υπέβαλα και που κατά την άποψή μου επιφέρουν θετικές αλλαγές στο κείμενο. Νομίζω ότι θα πρέπει να υιοθετήσουμε μια πάρα πολύ σκληρή προσέγγιση σε ό,τι αφορά την κατάχρηση της αγοράς ή των, ε, ε, ε, της πράξης χειραγώγησης. Γιατί σε συζητήσεις ε, που είχαμε ε, με τους ε, ρυθμιστές διαπιστώσαμε ότι τους απασχολεί το η αύξηση των ενδεχομένου για κατάχρηση της αγοράς. Βεβαίως ρυθμίζουμε τις αγορές και κατά συνέπεια υπάρχει η άποψη ότι θα υπάρχει ένας ακόμα μεγαλύτερος ε, πειρασμός ε, για χειραγώγηση των χωρών. Σε κάθε περίπτωση συμφωνούμε ότι θα πρέπει να είναι πάρα πολύ σκληρή η προσέγγιση μας. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονό ότι η Επιτροπή υπέβαλε αυτή την πρόταση. Αυτό που θα ήθελα να κάνω το σύντομο χρονικό διάστημα που έχω στη διάθεσή μου είναι να δούμε τις τροπολογίες και να ζητήσω τους σχέδους εισηγητής και τους εσείς και τους συναδέλφους να μιλήσουν για τις τροπολογίες θα γίνει μια συνάντηση και εισηγητών. Θα ήθελα να πω ευθύ εξ αρχή ότι προσπάθησα να ευθυγραμμίσω το χρονοδιάγραμμά μου με αυτό του κυρίου Φέρμπορ, γιατί οτιδήποτε κάνουμε στον κανονισμό αυτό που αφορά την ρύθμιση τη αγορά εξαρτάται από την πρόταση MIFID. Και κατά συνέπεια θέλουμε να γίνει σταδιακά συμφώνησα με τον κύριο Φέρμπερ ότι μερικές από τις τροπολογίες μου ενδεχομένω θα ενταχθούν καλύτερα στη δική του οδηγία. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ καλή και στενή συνεργασία. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε ορισμένους από τους τομείς όπου υπευλήθησαν τροπολογίες. Άρθρο 5 για τους οριμούς. Ε, σε ό,τι αφορά του ορισμούς. Μερικοί συνάδελφοι προσέθεσαν τροπολογίες σε ό,τι αφορά την αλλαγή των πρακτικών της αγοράς, των παραγόγων ε, ή της ε, διανομής. Υπάρχουν μερικές ε, αρκετές τροπολογίες εδώ και θα πρέπει να πω τη εξ αρχής ότι δεν έχω πρόβλημα για τροπολογίες που έχουν σχέση με τις πρακτικές της αγοράς. Νομίζω ότι είναι λογικό να τις εντάξουμε. Η κυρία Γκουλάντα αναφέρθηκε στον ορισμό των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Σε πρώτη ματιά δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Θα ήθελα να ακούσω και την άποψη των συναδέλφων. Μετά είχαμε... Ο κύριος Σμίτ επέφερε ορισμένε αλλαγέ ό,τι αφορά τον ορισμό του spot market. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρη για το θέμα αυτό. Θα ήθελα να το κοιτάξω με μεγαλύτερη προσοχή. Τι νόημα έχει το να αλλάξουμε τον ορισμό του spot market και να δω και τι επιπτώσεις έχει και αλλού. Έγινε και πάλι μια αναφορά στις φήμες που κυκλοφορούν και στον ορισμό, τον τρόπο που ε, ορίζονται. Θα πρέπει να ζητήσουμε από τις ρυθμιστικές αρχές να ορίσουν τι σημαίνουν φήμες για μια συγκεκριμένη αγορά ε, επίση έγινε μια αναφορά και στην σημαντική διανομή και στον ορισμό τη. Ενδεχομένω θα πρέπει να ελέγξουμε αυτές τις τροπολογίες γιατί θα μπορούσαν να βελτιώσουν το τελικό κείμενο. Αναφέρθηκα στις πράξεις κατεξοδησιοδότηση, ε, όταν υπάρχει κατάχρηση πρακτικών. Δεν υπήρχαν τροπολογίες ε, για αυτά, αλλά αυτά προσετέθησαν στην αρχική πρόταση Επιτροπή. Μετά είχαμε ένα αναφιλεγόμενο τομέα που αφορούσε τις, ε, τα πρόσωπα που κατέχουν επιστημονικέ πληροφορίε. Οι τροπολογίε αφορούσαν τις κατευθυντηρίους γραμμές ΕΣΜΑΝ, και τα ρυθμιστικά πρότυπα έσμα που θα πρέπει να αποκαλύπτονται στις αγορές παραγόγων. Με αυτόν τον τρόπο διαγράφεται η αναφορά στις σχετικές πληροφορίες. Ε, Θα πρέπει να πω ότι στο σχέδιο έκθεσης τροποποίησα το άρθρο 6 για να αναφερθώ στις επιπτώσεις που ε, έχουν στην αγορά των παραγόγων. Θα ήθελα λοιπόν να υπάρξει ένας καλύτερος ορισμός εδώ. Σε ό,τι αφορά το θέμα των σχετικών πληροφοριών και των εμπιστευτικών πληροφοριών, είμαι πεπισμένη ότι έχω καταφέρει να τα εξισορροπήσω. Δεν νομίζω ότι η διαγραφή είναι ο καλύτερος τρόπος γιατί είναι σαφές ότι θα θέλουν οι ρυθμιστές να ορίζουν τις σχετικές πληροφορίες. Θα προσπαθήσω όμως να δώσω στους συμμετέχοντες στην αγορά περισσότερα στοιχεία σχετικά με το τι θα μπορούσαν να αναμένουν. Αν υπάρχει μια εναλλακτική διατύπωση που θα μπορούσε να επιτύχει καλύτερα αυτό το στόχο, θα πρέπει να το εξετάσουμε. Είπα όμω ευθύ εξ αρχή ότι δεν ήμουν υπέρ του να διαγραφεί αυτό το θέμα για την ε, σχετική πληροφόρηση. Υπάρχουν άτομα που εμπλέκονται ε, έχουν εμπιστευτικές ε, πληροφορίες. Ο, παρόν όμως δεν τους συμπεριλαμβάνει και γι' αυτό το λόγο δεν ε, διώκονται. Γι' αυτό το λόγο μας ζητήθηκε να συμπεριλάβουμε αυτό το θέμα του σχετικού. Θα προσπαθήσω να το ορίσω, ενδεχομένως θα χρειαστεί περαιτέρω ενασχόληση. Είμαι κατά της ιδέας ε, του να το διαγράψουμε. Γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν θα μπορούν πλέον να ξεφεύγουν άτομα για απλά και μόνο γιατί δεν υπάρχει ένα σωστός ορισμός. Επίσης υπευλήθησα μερικέ τροπολογίες από ε, ένα συναδελφό μου ο οποίος υποστηρίζει το ζήτημα αυτό. Όπως σας είπα προσπάθησα να βρω ένα συμβιβασμό για να έχω τη βεβαιότητα ότι έχουμε το σωστό ορισμό που θα καλύψει το θέμα. Ε, ένας ε, ορισμός του λογικού επενδυτή. Με απασχολεί λίγο το θέμα ότι αυτό ξεπερνάει τον ορισμό αυτόν Ορισμένοι συνάδελφοι υπέβαλαν τροπολογίες ο κύριο Σμιτ, η κυρία ε, Λίμπε. Το θέμα είναι ότι αν κάποιος ε, καταδικαστεί για απάτη ο ορισμός αυτός δεν θα μπορούσε να βοηθήσει. Βεβαίως με χαρά θα το κοίταζα λεπτομερέστερα για να μπορέσω μαζί με τα μέλη να βρω ένα τρόπο για να καλύψω το ζήτημα. Οι άλλες απολογίες στο άρθρο 7 και 8 που αφορούν τη χειραγώγηση της αγοράς. Έκανα επιπλέον τροπολογίες μετά από τη συζήτηση με ρυθμιστές θα πρέπει να συμπεριλάβουμε το inside dealing με βάση συστάσει. Η, η σύσταση επιτροπής απαγορεύει από κάποιον να συστήσει με βάση εμπιστευτικέ πληροφορίες και να διαπραγματευτεί ε, αξίες. Παρόλα αυτά, δεν συμπεριλαμβάνεται κάποιο ο οποίο δρά με βάση αυτό το κίνητρο ή τη σύσταση. Καλύπτει κάποιον ο οποίο έχει εμπιστευτικέ πληροφορίε, αλλά όχι άτομα που βασίζονται σε αυτέ. Και αυτό είναι κάτι που, ένα παραθυράκι που θα πρέπει να κλείσουμε. Και οι δύο δραστηριότητε, κάποιο που έχει εμπιστευτικέ πληροφορίε και κάποιο ο οποίο ενημερώνεται από κάποιον που έχει εμπιστευτικέ πληροφορίε, θα πρέπει να καλυφθούν. Υπάρχουν ιδιαίτερα πολύπλοκα. Ε, μέσα πολλές φορές προσλαμβάνονται άτομα για τα οποία κάνουν συστάσεις και με βάση αυτό μπορούν να ε, κερδίσουν. Έκανα λοιπόν, ε, έχοντας στο νου ε, την τροπολογία, έχοντας στο νου μου το συγκεκριμένο αυτό σημείο. Είναι σαφές από τα πρακτικά παραδείγματα που μας έδωσαν οι ρυθμιστές ότι αυτοί που βασίζονται σε έναν ε, ε υπενιγμό κινούνται στην ουσία στο ίδιο επίπεδο και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με τον ίδιο τρόπο. Ο Συνάδελφο Σίμπερντ υπέβαλε τροπολογίε που ήταν παρεμφερεί. Τα μέλη υπέρευαλαν τροπολογίε για καταστάσεις οι οποίες δεν ταξινομούνται ως εμπιστευτικές πληροφορίες ε, που αφορούν μειοδοτικούς διαγωνισμούς, για παράδειγμα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε την κατα... τις καταστάσεις όπου δεν υπάρχουν περιπτώσεις διάθεσης εμπιστευτικών πληροφοριών. Οι τροπολογίες που κατατέθησαν ήταν πολύ ε, λογικές. Η κυρία Πετακάμνη υπέβαλε μια τροπολογία, μια λογική τροπολογία και εδώ παρόλα αυτά το πρόβλημα είναι ότι ο κύριος Γκούλαρντ ε, αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα. Νομίζω ότι θα πρέπει να το κοιτάξουμε λεπτομερέστερα. Ίσως είναι το πρόβλημα με το γαλλικό δίκαιο. Συνεπώ θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε μία λύση σε αυτό. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να ορίσουμε το τι εννοούμε προσπάθεια. Αυτό το αναφέρει και η Επιτροπή και το Συμβούλιο. Προσπάθειες συμπεριλήφθησαν και στις προηγούμενες οδηγίες και συνεπώς δεν θα πρέπει να αποδυναμώσουμε αυτό τον κανονισμό. Θα πρέπει τουλάχιστον να έχει όσα είχε και προηγούμενος. Στο άρθρο 8, χειραγώγηση της αγοράς. Έχω μερικές χρήσιμες πληροφορίες που υπευλήθησαν εδώ από τους κυρίου Παδεκάνε, Φερέρα και μία τροπολογία από την κυρία Σουίμπονση, η οποία συμπεριλαμβάνει ε, το ε, πολύ σε τεχνικό επίπεδο. Είχα κάποια ανατροφοδότηση από τους ενδιαφερόμενους σχετικά με το θέμα της δημιουργίας τιμών σε ένα μη φυσιολογικό επίπεδο. Υπάρχει και μια καινούργια παράγραφος για πληροφορίες που θα πρέπει να δημοσιοποιούνται. Νομίζω ότι θα πρέπει να ασχοληθεί ασχοληθούμε με αυτό το θέμα της επιχειρούμενης ε, κατάχρησης της αγοράς που θα πρέπει να διαγραφεί. Θα πρέπει να έχουμε τη βεβαιότητα ότι υπάρχει η ακαιρεότητα της αγοράς. Αν κοιτάξουμε το άρθρο 13, insider list, πρόσωπα που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες, είναι πολύ χρήσιμα εργαλεία για τις αρμόδιες αρχές. Οι συνάδελφοι θα θυμούνται ότι στην πρώτη παρουσίαση της έκθεσης διέγραψα την αναφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συμφωνώ ότι γενικά θα πρέπει να αναζητήσουμε τρόπους για να, να μειώσουμε το διοικητικό δο, ε, ε, ε, βάρος. Σε περίπτωση όμως της κατάχρησης αγοράς θα πρέπει να υπάρξει μία εξαίρεση είναι μια θεμελιώδης αρχή για την προστασία των επενδυτών. Όλες οι αγορές θα πρέπει να εφαρμόζουν τους ίδιους κανόνες. Ε, κοιτώντας το αυτό με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, βλέπω ότι στη Φιλανδία το 99% είναι μικρές επιχειρήσεις, άρα υπάρχει το 99% που θα πρέπει να καλύπτεται από τον κανονισμό. Επιπλέον, το ανέφερα και την τελευταία φορά, υπάρχει μια τάση προς αυτό που ονομάζουμε boutique ε, ε, traders, αυτοί δηλαδή είναι ε, που έχουν πολύ μικρούς, ε, λίγους πελάτες, όχι μπορεί να είναι μικρός αριθμός ακόμα και αν είναι μικρή επιχείρηση. Και επίσης υπάρχουν και μεγάλες εταιρείες όπως η JP Morgan, η Goldman Sachs και η Τράπεζα της Αμερικές λένε ότι είναι και οι ίδιες μπουτίκ εταιρείες και πηγαίνουν στον κλάδο των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εγώ το διέγραψα αυτό. Ε, το, ε, νομίζω ότι ως συμβεβασμό θα μπορούσαμε να διευκολύνουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο να πληρούν αυτούς, αυτές τις απαιτήσεις. Στις συζητήσεις Ε, με την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, αν δείτε το έγγραφό τους, λέει εκεί ότι οι κανόνες ε, για τις συναλλαγές προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες είναι μία υποχρέωση που θέλουν οι εταιρείες να έχουν. Δεν ε, εξυπηρετεί πιο στόχο λοιπόν να αφαιρούμε υποχρεώσεις που οι ίδιες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θέλουν να έχουν. Απλώς μπορούμε να τις διευκολύνουμε, να κάνουμε τα πράγματα πιο εύκολα, να τους δώσουμε μια ε, λίστα με τα πρόσωπα που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες στο διαδίκτυο για να μην έχουν περισσότερη δουλειά να κάνουν στο να τους βρίσκουν. Ο βασικός ε, ε, ε, λόγος είναι ότι αυτά τα σχέδια Ponzi και οι boutiques είναι υπηρεσίες ιδιαίτερα προσωπικές θα έλεγα. Άλλα μέλη επίσης, άλλοι βουλευτές κατέθεσαν πολύ καλές τροπολογίες όπως η απέτηση να ορίζονται από την ΕΑΚΑ τα στοιχεία και όχι από την Κομισιόν. Η πρόταση της Κομισιόν δεν δίνει χρόνο, αλλά ε, αφήνει στις ε, πράξεις κατά εξουσιοδότηση να αποφασίσουν. Άρα η ΕΑΚΑ θα πρέπει να δώσει κάποιες, ΕΚΑ θα πρέπει να δώσει τις λεπτομέρειες. Επίσης ε, υπάρχουν υποχρεώσεις ρυθμιστικές και υπάρχουν τροπολογίες για αυτές, τροπολογίες που υποστηρίζουν ε, τη διαγραφή της εξαίρεσης για τις μικρομεσαίες ε, λένε ότι πρέπει οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, να βοηθηθούν στο να κατανοήσουν τους κανόνες και να μην τους παραβαίνουν επειδή δεν τους κατανοούν. Στο άρθρο 14 τώρα έσβησα το κατόφλι για την αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τις συναλλαγές. Ε, η αποκάλυψη πληροφοριών θα πρέπει να γίνεται μέσα σε δύο εργάσιμες μέρες από την ημέρα της συναλλαγής λαϊκών μισιών. Αν θυμάστε συνάδελφοι, είχα και εγώ ε, βάλει αυτή την ιδέα ενός παραθύρου συναλλαγών μέσα στο οποίο θα πρέπει να μπορούν να γίνονται οι συναλλαγές. Όμως ε, μου είπανε οι ενδιαφερόμενοι ότι ε, είναι καλύτερο να μπορούν εντός ενός παραθύρου να ε, κάνουν τις συναλλαγές τους παρά εκτός και γι' αυτό μάλλον πρέπει να δουλέψουμε λίγο παραπάνω αυτή την πρόταση. Άτυπα η Κομισιόν μου είπε ότι τους αρέσει αυτή η ιδέα του να υπάρχει αυτό το παράθυρο και αν θυμάστε συνάδελφοι προσπαθήσαμε να δούμε κάποια πρακτικά ε, παραδείγματα εταιριών που έκαναν τις συναλλαγές τους, ε, πούλησαν δηλαδή τις μετοχές τους, λίγο πριν βγουν τα νούμερα και ε, είχαν 300.000 και 400.000 λίρες ως αντάλλαγμα και υπήρχαν και άλλες εταιρείες που δεν μπόρεσαν επειδή δεν είχαν εμπιστευτικές πληροφορίες και έχασαν την ευκαιρία. Άρα πρέπει ε, να υπάρχει στο σύστημα κάποια πρόβλεψη και γι' αυτό. Η καταγραφή των ε, υποχρεώσεων για τις ε, συναλλαγές, η καταγραφή των συναλλαγών των managers είναι κάτι που θα πρέπει να δίνεται γιατί οι manager μας δείχνουν έτσι τι σκέφτονται για τις τιμές ε, θέλουμε να έχουμε διαφανείς αγορές, θέλουμε να έχουμε εμπιστοσύνη των επενδυτών. Η Κομισιόν επίσης προτείνει οποιαδήποτε συναλλαγή ε, γίνεται ε, από κάποιον να δηλώνεται στις δημόσιες αρχές όταν υπάρχει κάποια ε, πολύ ενός μάνατζερ. Είναι λογικό μέσα σε δύο ημέρες να γίνεται η αποκάλυψη των πληροφοριών. Δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ε, κατόφλι για να κλείνουν. Ε, αν δεν, μπορεί κανείς, αν δεν έχει κανείς κάτι να κρύψει, γιατί να μην αποκαλύψει ποιες είναι οι συναλλαγές. Επίσης με ανησυχεί λίγο, αλλά ίσως οι συνάδελφοι μπορούν να μου πούνε και να μου δικαιολογήσουν γιατί σε κάποιες περιπτώσεις ζήτησαν μεγαλύτερο κατόφλι. Αρχικά στην οδηγία είχαμε νομίζω 5.000 ε, ε, στην οδηγία της Κομισιόν ε, και στην άλλη οδηγία αυξήθηκε στις 20.000. Τώρα οι συνάδελφοι βάλανε 50.000 και έχουν βάλει και μία ρήτρα reset που δεν ξέρω ποια είναι η χρησιμότητά της. Ο κύριος Κανφάντ διέγραψε το κατόφλι. Επίσης ε, έβαλε ένα παράθυρο μιας εβδομάδας ε, μετά από την ε, δημοσίευση των ετήσιων εκθέσεων. Η κυρία Κένφκανς διατήρησε το window, αλλά πρέπει το παράθυρο, αλλά πρέπει να το ορίζει η ΕΚΑ. Νομίζω ότι και εδώ μπορούμε να βρούμε μια σωστή λύση, έναν καλό συμβιβασμό μεταξύ των τροπολογιών. Τώρα στο άρθρο 17 έχουμε τις ε, αρμόδιες αρχές. Ε, υπάρχουν τροπολογίες ε, που κατατέθηκαν και από το Συμβούλιο, οι οποίες διασφαλίζουν ώστε οι κατάλληλες, οι αρμόδιες υπηρεσίες να έχουν τα εργαλεία για να αποφεύγουν την κατάχρηση της αγοράς λίγο πιο αργά μπορεί η ομιλήτρια για να προλαβαίνουν οι διερμηνείς. Υπήρχε μεγάλη συμφωνία στις τροπολογίες έτσι ώστε να έχουν τα εργαλεία οι αρχές για να μπορέσουν να ε, παγώσουν ας πούμε κεφάλαια, ε, να διακόψουν ε, προσωρινά συναλλαγές ώστε να ρυθμίσουν να ελέγχουν τέτοια ζητήματα. Να δημεύσουν επίσης. Ένα άλλο θέμα που ε, φύγει η MIFID και γίνεται συζήτηση ε, και για το οποίο πρέπει να υπάρχει συνέπεια και συνοχή είναι το ακόλουθο. Θα πρέπει να ε, διασφαλίσουμε την διασυνοριακή εποπτεία. Όπως είπα, ε, στο περιβάλλον που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα μετοχικά προϊόντα είναι ε, δύσκολο κανείς διασυνοριακά να ανοιχνεύσει την κατάχρηση της αγοράς. Αυτό που έκανα εγώ ήταν να εισάγω ε, τροπολογίες για τις αρμόδες αρχές των πιο σχετικών αγορών σε επίπεδο ρευστότητας για χρηματοπιστωτικά εργαλεία έτσι ώστε ε, να ε, μπορεί κανείς να γνωρίζει για όλους τους πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης στοιχεία. Ξέρω ότι οι συνάδελφοι θα πούνε ότι είναι πολλά ε, αυτά τα στοιχεία, αλλά υπάρχει, ε, φαίνεται μια τάση υποστήριξης αυτών των προτάσεων μου. Κάποιες από τις τροπολογίες ζητούν από την αρμόδια αρχή ε, της αγοράς όπου έγινε πρώτη έκδοση να είναι υπεύθυνη για την εποπτεία. Η κυρία Πετκάνεν και ο κύριος Κλίνς ε, κατέθεσαν τέτοιες τροπολογίες, όμως ε, σε αυτές ε, αναφέρεται ε, ότι θα πρέπει να είναι οι αρχές που γίνεται η πρώτη έκδοση ο κύριος ε, Σμιτ ανέφερε το θέμα της εποπτείας και πάλι εκεί που ε, το χρεόγραφο για πρώτη φορά εκδίδεται. Νομίζω, συνάδελφοι, ότι για αυτό το θέμα πρέπει να συζητήσουμε πάρα πολύ στις κοιόδεις συναντήσεις μας ε, πριν βγάλουμε τελικό συμπέρασμα. Νομίζω ότι οι ρυθμιστές σε διασυνοριακό επίπεδο θα ήταν πιο αποδοτικοί αν είχαμε την αγορά όπου υπάρχει μεγαλύτερη ρευστότητα και αυτό θα μπορεί να το δούμε μέσα από το τρέμ, από τον ε, μηχανισμό ε, της ε, καταγραφής των αγορών. Και ε, σύμφωνα με το MIFID ε, λέει ότι η ΕΚΑ θα είναι αυτή που θα ορίζει ποια είναι η πιο ρευστή αγορά. Έτσι θα μπορούμε μέσα από την εποπτεία να πετύχουμε το στόχο μας, όμως αυτό θα το συζητήσουμε με τους συναδέλφους, γιατί έχουμε διαφορετικά επιχειρήματα για διάφορους θέσεις. Ποια θα είναι η πρώτη αγορά ή η πιο ρευστή αγορά με τη μεγαλύτερη ρευστότητα. Ε, καταχρηστική χρήση του ε, ε, στο ε, order book ε, το είπα ξεχάθαρα στους ε, συναδέλφους ότι θέλω να υπάρχουν μέτρα αποτροπής ε, ώστε να μην γίνονται καταχρήσεις. Ε, στην έκθεσή μου αναφέρω την υποχρέωση των χειριστών να αποφεύγουν την κατάχρηση των βιβλίων ετολών θα πρέπει να δούμε από ποιο σημείο και μετά θα πρέπει όποιο συμμετέχει στην αγορά να πληρώνει κάποιο τέλος. Στη ΜΥΦΙΤ πρέπει να έχουμε τις ίδιες απόψεις, αλλά δεν ήθελα να γίνει η συζήτηση μέσα στα πλαίσια του κανονισμού. Ε, ήθελα να γίνει συζήτηση μέσα στα πλαίσια του κανονισμού για την κατάχρηση της αγοράς, γιατί μιλάμε για κατάχρηση και νομίζω ότι πρέπει να το συζητήσουμε ε, ε, και να διασφαλίσουμε η ΜΥΦΙΤ να έχει ε, κάποια στοιχεία γι' αυτό. Υπάρχουν επίσης ε, τα ratios ε, που πρότειναν πολλά μέλη, πάλι να ορίζονται από την ΕΚΑ. Χαίρομαι που κατέθεσαν εναλλακτικέ απόψει οι συνάδελφοι, αλλά και πάλι πρέπει ω και να συζητήσουμε πριν φτάσουμε σε τελικό συμπέρασμα. Όπω είπα προηγούμενα στη συζήτηση για τη ΜΥΦΙΤ. Ε, ο κύριος Γκέμπελς ε, θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί ε, να έχουμε αυτή την περίοδο κράτησης 500 εκατοστών του δευτερολέπτου. Όμως γενικά θα πρέπει να έχουμε μια συνεκτική μια συνέχεια μεταξύ της ΜΥΦΙΤ και της οδηγίας κατάχρησης της αγοράς. Τη όλους τους σκιώδες και να πω ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ώστε στη ΜΥΦΕΤ να υπάρχουν δυνατότητες ε, για αντιμετώπιση των στοιχείων που έχουν να κάνουν με κατάχρηση αγοράς. Να πάω τώρα στις κυρώσεις. Στο άρθρο 11. Εδώ έχουν εισαχθεί πάρα πολύ ε, σωστές τροπολογίες για να ε, καταγράφονται οι παραβιάσεις εκ μέρους αυτών οι οποίες ε, στις οποίες επιπίπτουν αυτοί που έχουν εμπιστευτικές πληροφορίες, είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν, όπως λέει ο κύριος Κλίνς, ε, οι διασφαλίσεις ότι θα επιβάλλονται κυρώσεις σε περίπτωση που υπάρχουν αξιόπινες πράκλες. Και επίσης οι ρυθμιστικές αρχές θα μπορούν ε, να εισαγάγουν ε, περιόδους ε, κυρώσεων περισσο, ίσως και ως δύο χρόνια. Ο κύριος ε, Κανφέ, ο κύριος Σμίτ, ο κύριος ε, επίση έχουν καταθέσει τροπολογίε. Θα πρέπει να βρούμε όμως εμείς μια κοινή λύση, διότι άλλοι συνάδελφοι προτείνουν ε, μικρότερες, άλλες μεγαλύτερες κυρώσεις. Επίσης, για το θέμα της ε, αναφοράς των παραβιάσεων, πολλοί συνάδελφοι κατέθεσαν τροπολογίες. Ο κύριος Σμιτ κατέθεσε μία τροπολογία επίσης για τα χρηματοπιστωτικά κέντρα και ε, εδώ πρέπει να πω ότι έχουμε να κάνουμε με μία εναλλακτική λύση η οποία προσφέρεται και όχι υποχρέωση από την οδηγία. Επίσης, όσον αφορά την ε, στρατηγική που πρέπει να έχουμε όλοι, όπως είπε και η κυρία Μπόλ στην τροπολογία της, κατά των ε, ε, απάτης, θα πρέπει να δούμε γιατί ακριβώς μιλάει. Για μια ενιαία στρατηγική κατά τις απάτες ή εκεί όπου χρειάζεται θα πρέπει με περισσότερε λεπτομέρειε να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Επίσης, το άρθρο 11. Έχουμε ε, τροπολογίες που ζητούν από την ΕΚΑ και τις ε, ε εθνικές αρχές να ασχοληθούν με τα θέματα αυτά της ε, ε, προστασίας των ατόμων τα οποία έχουν καταθέσει ε, τέτοιου είδους τροπολογίες. Πολλές φορές πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν συνάδελφοι, οι οποίοι, ε, όπως λένε οι συνάδελφοι, υπάρχουν άτομα τα οποία δεν ε, θέλουν να, να διασφαλιστεί το ανώνυμο της καταγγελίας. Τώρα, τροπολογίες 4 42. αλλά σταματήσω προς το παρόν να ακούσω τις απόψεις και θα επανέλθω στα θέματα των συγχωνεύσεων μετά. Ευχαριστώ. Ε, έχουμε λίγο χρόνο ακόμη πριν να αρχίσουμε την ε, συζήτηση για τον προπολογισμό. Θα δώσω το λόγο σου και όσοι ΣΥΡΠΑ πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ συνεκτική και σύντομη. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την επικοδομητική συνεργασία και την εμπεριστατωμένη δουλειά της που έκανε για την έκθεση αυτή. Και όντως νομίζω ότι εδώ μπορούμε να συζητήσουμε και να καταλήξουμε στα κύρια θέματα σε συμβιβασμούς. Πρώτα απ' όλα, πεδίο εφαρμογής, το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει παντού η ίδια ρύθμιση, οι ίδιοι κανόνες για όλους, ώστε να καλύπτονται από την κανονισμό. Όσον αφορά τις εμπιστευτικές ε, πληροφορίες, νομίζω ότι καλύφθηκε λεπτομεριακά το θέμα. Είμαι υπέρ του να υπάρχουν τέτοιου είδους πληροφορίες, διότι όλοι ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να οριστούν οι περιπτώσεις στις οποίες όντως ε, τέτοιου είδους πληροφορίες χρησιμοποιούνται αρνητικά. Επίσης, θα πρέπει όλες αυτές οι πληροφορίες που μπορούν να γίνουν αποδεκτές ώστε να υπάρχει μια σωστή συμπεριφορά θα πρέπει να καθοριστούν ότι υπάρχουν κάποιες συμπεριφορές που είναι απαράδεκτες, δεν μπορούν να γίνουν ε, αποδεκτές. Τώρα, όσον αφορά τις αλγοριθμικές και υψηλή συχνότητα συναλλαγές, είναι κάτι το οποίο το συζητήσαμε μεταξύ μας διεξοδικά. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές ε, καταχρήσεις στην αγορά. Δεν είναι εύκολο να το χειριστούμε το θέμα. Κατά την άποψή μας και κατά τη δική μου ε, άποψη, θα πρέπει να δούμε πώς έχει η ε, δομή, πώς διαμορφώνεται η δομή των ε, προμηθειών για να μην έχουμε προβλήματα. Τώρα, όσον αφορά την χειραγώγηση των αγορών, νομίζω ότι θα πρέπει εδώ να έχουμε γενικέ αρχέ, αλλά νομίζω ότι μπορεί να οδηγηθούμε σε, τέτοι... σε κάποιες αγορές, σε κάποια κρατημέλη όπως την Γαλλία σε τέτοιες πρακτικές. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει νομική κάλυψη και νομική ασφάλεια στο τι ακριβώς είναι αυτό. Νομίζω ότι είναι σημαντικό λοιπόν να το συμπεριλάβουμε εδώ. Ακούσαμε ε, επίσης να μιλάτε για τις ε, μιμιές, για τις μιμιέ, διότι είπατε ότι πολλές περιπτώσεις δεν θέλουν να θεωρούνται δεύτερες κατηγορίες δεδομένου ότι δεν αποτελούν το κύριο ενδιαφέρον εκ μέρους των ε, επενδυτών. Μιλήσατε τώρα επίσης για τις περίφημες boutique ε, εταιρείε όσον αφορά τους διαχειριστές. Είπατε ότι υπάρχουν αυτά τα παραθυράκια για τις ε, συναλλαγές. Θα ήθελα απλώ να πω ότι ούτως ή άλλως οι διαχειριστές σχεδόν πάντα έχουν τέτοιου είδους επιστατικές προφορές εξαιτία της δραστηριότητας που αναπτύσσουν. Άρα, εάν δεν υπάρχει περαιτέρω μεν, δεν θα επιληθεί το πρόβλημα. και θα πρέπει να το λύσουμε αυτό διότι είναι σημαντικό μέρος. Όσον αφορά τα κατόφλια, είπατε ότι δεν γίνεται τίποτα μέχρι τις 2.000. Ε, αυτό δεν είναι τόσο σημαντικό. Διότι οι συναλλαγές συνήθως υπερβαίνουν τι 2.000. Και είναι και θέμα γραφειοκρατίας το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Κατά την άποψή μου πάμε προς την σωστή κατεύθυνση όσον αφορά αυτές τις ε, εμπιστευτικές πληροφορίες με τη φάση των οποίων ενεργούν ορισμένα άτομα και τελευταία παρατήρηση εποπτεία των αγορών. Κατέθεσα τροπολογίες για τις ε, αρμόδιες αρχές και μίλησα για τις ε, ε, primary list. Δεδομένου ότι κάποιοι έχουν εκεί τις κατάλληλες πληροφορίες για κάποια εταιρεία και μπορούν να έχουν και άμεση πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Από ότι οι αγορές για θέματα ρευστότητος. Αλλά όλα αυτά τα θέματα θα συζητήσουμε, να τα συζητούμε στην συνάντηση των σκιωδών. Ο Γουλφ Κλίντ. Ευχαριστώ. κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι μπορούμε, ε, δεν πρέπει να υποτίμησουμε τη σημασία αυτού του θέματος στην Νέα Υόρκη τις τελευταίες εβδομάδες είδαμε πόσο, σημαντικά, πόσο μεγάλη σημασία δίνουν οι Αμερικάνοι στις κυρώσεις για πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες. Γι' αυτό θα πρέπει ε, να διασφαλίσουμε με την εφαρμογή ε, αυτής της ε, οδηγίας να μπορούμε οι ευρωπαϊκές αγορές να παραμένουν ελκυστικές διεθνώς. Θα πρέπει λοιπόν η εφαρμογή να μην είναι έτσι τυχαία ε, και κατακαιρματισμένη. Ταυτόχρονα υπάρχει μια σειρά ζητημάτων που παραμένουν ανοιχτά όσον αφορά στους στόχους. Καταρχάς ε, θεωρώ ότι η οδηγία από το 2003 ε, αναφέρει ε, έναν ορισμό για αυτές τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες. Ε, για μια άλλη εταιρεία ας πούμε και χρησιμοποιούν αυτές ε, τις ε, πληροφορίες με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν τον έλεγχο αυτής της εταιρεία και σε αυτή την έκθεση τώρα ε, δεν αναφέρεται ξεκάθαρα αυτή η περίπτωση. Άρα ισχύει αυτό που εγγράφεται στην οδηγία του 2003 ή ισχύει με άλλη μορφή, ξέρω εγώ ή όχι. Για την ε, MIFID λοιπόν, ε, για την λίστα των προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες δεν χρειαζόμαστε εξαιρέσεις. Πρέπει όλα να περιλαμβάνονται μικρές, μεγάλες επιχειρήσεις, έτσι ε, ώστε να μην υπάρχουν διαφορές. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ε, το κόστος ε, για τις επιχειρήσεις θα αντιμετωπίζεται Γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα ενιαίο, μια ενιαία και εναρμονισμένη πρόταση για αυτές τις λίστες. Όσον αφορά τον ορισμό των εμπιστευτικών πληροφοριών, ε, το Συμβούλιο ε, έχει σβήσει αυτό το άρθρο, όχι γιατί το θεωρεί ότι δεν είναι χρήσιμο, αλλά επειδή χρειάζεται πολύ μεγάλη επεξεργασία. Θα πρέπει λοιπόν στην πράξη να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια πολύ καλή επεξεργασία αυτού του ορισμού. direct dealings. Ε, νομίζω ότι όπως ε, φαίνεται ότι αυτό δεν συμβαίνει τίποτα άλλο παρά το γεγονός ότι όταν φτάσουμε στο 2020 στη 20.000 μάλλον ε, θα πρέπει να αναφέρεται ότι ο Τάδε ή ο Δίνα έχει κάνει 20.000 συναλλαγές. Θα αποφεύγουμε Απλώς ε, να μην ε, γίνεται δήλωση για κάθε 500 ευρώ πώληση ή δήλωση. Τώρα, για την εποπτεία της αγοράς. Ε, ως τώρα δεν είχα καταλάβει γιατί θα πρέπει το IPO να θεωρείται σημείο για την εποπτεία τώρα. Όμως υπάρχει αυτό το εύλογο επιχείρημα του που είναι η αγορά με τη μεγαλύτερη ρευστότητα είναι ε, οι περισσότερες ε, εταιρείε ε, αυτού του είδους, οι περισσότερες συναλλαγές αυτού του είδους γίνονται ίσως στο Λονδίνο. ίσως θα μπορούσε να είναι το Παρίσι ή κάποιες άλλες αγορές, αλλά βασικά είναι το Λονδίνο και ίσως να υπάρχουν και νέε αγορές στην Ανατολική Ευρώπη, οι οποίες δεν θα αντιμετωπίζονται με ίδιο τρόπο. Δεν θα ήθελα επίσης να έχουμε ρυθμίσεις οι οποίες να οδηγούν σε μια κουλτούρα ε, κατασκοπίας ας πούμε. Είμαι πολύ προσεκτικός, έχω αυτές τις ε, αναστολές. Ε, υπάρχουν οι διοικητικές κυρώσεις, ε, εντάξει μπορούμε να έχουμε, δεν υπάρχει θέμα σε αυτό, αλλά 10% του τζίρου, του ετήσιου τζίρου, για κάποιες εταιρείε αυτό θα τις οδηγήσει στην καταστροφή. Το 10% του τζίρου ε, ίσως θα ήταν σωστό να πάει στα κέρδη. Είναι ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να το λύσουμε. Και η συνεργασία με την ΕΑΚΑ είναι σημαντική σε αυτό το σημείο. Για τη δήλωση των ε, συναλλαγών μέσα σε τρεις μέρες ε, το θεωρώ ότι ε, γίνεται. Σε πολλές φάσεις της ζωής μου ήμουνα μη εκτελεστικός ε, διευθυντής και μπορούσα να κάνω τη δήλωση μέσα σε μία μέρα. δεν ξέρω γιατί είναι τόσο προβληματικό, αλλά ίσως σε κάποιες χώρες να υπάρχουν άλλες διαδικασίες, να υπάρχει ανάγκη για μια επίσημη επικύρωση πριν γίνει αυτή η δήλωση. Δεν ξέρω, αυτά είναι σχετικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά μας πιέζει ο χρόνος. Δεν μπορούμε να αναβάλουμε τη συζήτηση για τον προπολογισμό. Δεν ξέρω, Κέι, να δώσουμε αυτή τη φορά σε σένα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, γιατί ήδη ήταν ε, μεγάλο εγχείρημα το να εξετάσει και τα δύο αυτά θέματα. Θα ήθελα να επικεντρώσω την προσοχή μου σε ορισμένα θέματα. Τονίζουμε ότι η προσπάθεια χειραγώγησης της αγοράς είναι το ίδιο πράγμα με μια επιτυχή χειραγώγηση της αγοράς. Νομίζω ότι αυτό θα μπορέσουμε να το κάνουμε και θα πρέπει να το τονίσουμε όπως εξάλλου προσπάθησαν να κάνουν πολλοί συνάδελφοι. Σαφώς υποστηρίζω ότι αυτό είναι η πρόθεση όλων μας να εξισώσουμε την ε, επιδιωκόμενη με την πραγματοποιημένη χειραγώγηση της αγοράς. Νομίζω ότι θα πρέπει να εφαρμόσουμε μια προσεκτική πολιτική και είναι δύσκολο να γίνει αυτό. Και αυτό θα πρέπει να ισχύει για όλα τα επίπεδα, για όλες τις εταιρείε. Θα πρέπει να διακρίνουμε τις σχετικές εμπιστευτικές πληροφορίες σε σχέση με τις απαγορεύσεις που είναι μια ευρύτερη έννοια και ενδεχομένως θα, θα δημιουργήσουν αντικίνητρα σε πολλούς επενδυτές. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε μια ισορροπία, να δούμε τι απαιτείται εδώ. Με προβλημάτισε το άρθρο 4α που έχουμε τις ε, πρακτικές της αγοράς. Θα έλεγα ότι αρχίζουμε να εξαλείφουμε τις ε, ε, τρέχουσες πρακτικές της αγοράς ε, στις χώρες μέλη, ότι ενδεχομένως χρειάζεται μία σειρά από αρχές θα ήθελα να γνωρίζω τι είδου εθνικές εξαιρέσεις θα μπορούσαν να ε, συμπεριληφθούν σε αυτές τις ε, αποδεκτές πρακτικές της αγοράς όπως εμφαρίζονται στο κείμενο. Η εποπτεία της αγοράς. Υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ, διάβασα προσεκτικά το κείμενο. Προτιμάω την αρχική πρόταση Κάπως με απασχολεί το θέμα του να επιλέξουμε ένα και μοναδικό σημείο που να είναι υπεύθυνο για την, ένα τόπο συναλλαγής που να είναι υπεύθυνο για την ε, εποπτεία. Δεν έχω την βεβαιότητα ότι θα μπορούσε να γίνει μία διάκριση σε ό,τι αφορά τον τόπο αυτών των συναλλαγών. Το θέμα είναι να δούμε πού βρίσκεται η ρευστότητα. Λίγο με προβληματίζει κατά πόσο θα μπορούσε να γίνει αυτή η διάκριση στα πλαίσια του ΜΥΦΙΔ. Νομίζω το ευρωπαϊκό μοντέλο του ΜΥΦΙΔ διαφέρει από το αμερικανικό εκεί στις πρωτογενείς αγορές υπάρχει και η εποπτεία, υπάρχει και ο κανονισμός, υπάρχουν ορισμένα βασικά θέματα εδώ. Δεν θα πρέπει όμως να μεταφέρουμε ένα αμερικανικό μοντέλο ε, στην Ευρώπη, γιατί το MIFID είναι ένα πολύ καλό, μια πολύ καλή βάση. Μπορώ να καταλάβω αυτό που είπε η Αρλίνα ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες. Αυτό που προσπαθήσαμε να τονίσουμε είναι ότι ε, πολλές φορές είναι θέμα γραφειοκρατίας. Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να τα διατηρήσουμε όλα αυτά. Χαίρομαι που η συγγήτρια προσπάθησε να βρει τρόπους για να μπορέσει να λειτουργήσει η αγορά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. θα πρέπει να διασφαλίσουμε την λειτουργία των αγορών στα πλαίσια του MIFID. Οι αγορές της ε, Σιγκαπούρης ε, έχουν στρέψει τα βλέμματα προς εδώ. έτσι ώστε να υπάρξει συμμόρφωση με την νομοθεσία που, είναι, ε, που αφορά την κατάχρηση των αγορών. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Θα πρέπει η αγορά ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να είναι μια βιώσιμη αγορά για όλη την Ευρώπη. Χαίρομαι ιδιαίτερα με την πλειοψηφία των όσων αναφέρονται σε αυτή την έκθεση και με χαρά θα περίμενα να ακούσω τα σχόλια από τον εισηγητή. Περιμένω λοιπόν τις επόμενες εβδομάδες να μας υποβληθεί το κείμενο συμβιβασμού. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας τονίσω ότι ο χρόνος μας πιέζει ότι κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την προσέγγιση της για το όλο θέμα, σε θέματα διαδικασίας και περιεχομένου. Θα ήθελα κάποια κύρια θέματα για μας να αρθρο Άρθρο 10α έχουμε προβλέψει κάτι για τις παραβάσεις και θέλουμε να υπάρχει ε, μεγαλύτερο πόσο ε, και αναλογία όχι 10 προς 1, 50 προς 1. Επίσης, πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει μία καλύτερη προσέγγιση σε σχέση με αυτούς οι οποίοι παρέχουν τέτοιου είδους πληροφορίες. Αντίθετα με αυτά που είπε ο Wall Cliff και κρίμα ε, που δεν είναι εδώ, πρέπει να πω ότι πολλές φορές ε, ε, to highlight with... τα παπαγαλάκια που επαναλαμβάνει πληροφορίες υπάρχουν σε όλες τις εταιρείε και θα πρέπει για να μην υπάρχουν καταχρήσεις να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στο ρόλο που παίζουν. Νομίζω ότι θα πρέπει εδώ κάτι να κάνει το Κοινοβούλιο. Τώρα, στο 11.2 νέο θέλουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει η υποχρέωση αναφοράς ε, ε, θεμάτων κατάχρησης εκ μέρους ανθρώπων που έχουν εμπιστευτικές ε, τροπολογίες. Στο 12, 2 και 3 λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει διευκρίνηση της ε, διαδικασίες που προβλέπεται όταν καθυστερείται η διάθεση πληροφοριών. Επίσης, θα πρέπει να προβλέψουμε κάτι για τις πληροφορίες οι οποίες δίδονται μετά από την δημοσίευση των τριμηνίων εξαμενίων εκθέσεων. Όσον αφορά το άρθρο 26.1 λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις ε, που να προβλέπουν προσωρινή μόνιμη απαγόρευση και δύο ετών ποινική κηρύση αν υπάρχει τέτοιο είδους πρόβλημα ε, παραβίασης των κανόνων της αγοράς εξαιτίας εμπιστευτικών πληροφοριών. Σε πολλές άλλες υποπαραγράφους και άρθρα, το άρθρο 26 επίσης, προβλέπουμε ενίσχυση του όλου συστήματος επιβολής ποινών. Τώρα, όσον αφορά τις τροπολογίες κάποιων συναδέλφων, Όλε Σμιτ, πρέπει να πω ότι δεν ε, ε, περιλαμβάνει τον ε, ορισμό ε, τη συμπεριφορά σε περίπτωση παραβίαση αγορά. Εμεί πιστεύουμε ότι αν μιλήσουμε μόνο για συμπεριφορά, δεν είμαστε πεπισμένοι ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι ε, το οποίο να μας καλύπτει νομικά. Οι Γκόζες, Πιτικάινεν και Μπερές θέλουν να διευκρινίσουν την ε, ε, θέσπιση κάποιων πρακτικών που είναι αποδεκτές σε κάποιες αγορές και νομίζω ότι αυτό είναι σωστό. Χαιρετίζουμε επίσης τροπολογίες που κατέθεσαν διάφορα μέλη για να εξασφαλιστεί ότι οι δημοσιογράφοι δεν ε, θα χρησιμοποιούν τέτοιου είδους πληροφορίες που αφορούν ε, την ε, κατάχρηση στην αγορά. Όσον αφορά αυτά τα Chinese walls, τα στεγανά πληροφόρησης, πιστεύουμε ότι δεν μπορούν να προστατεύσουν κάποιο. Έρθρο 7, παράγραφος 7. Θα πρέπει να διαγραφεί. Χαιρετίζουμε την τροπολογία 229 της εισηγητρίας που λέει ότι ε, παρά το γεγονό ότι κάποιος αποτυγχάνει να χειραγωγήσει τις αγορές, ε, θα πρέπει να είναι επιλήψιμη η πράξη του αυτού, παρόλο ότι θα αποτύχει. Επίσης, η ΕΚΑ θα πρέπει να ενημερώνει πάντα την κείμενη νομοθεσία και να λαμβάνει υπόψη τις νέες τεχνολογίες που μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ η Μαρίζα Ματιές. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την περιμπεριστατωμένη και σαφέστατη ανάλυση των θεμάτων που μας απασχολούν σε θέση με αυτή την οδηγία. Ξέρουμε ότι πρόκειται για νομοθεσία που απαιτεί μεγάλη ακρίβεια στους ορισμούς και μεγάλη διευκρίνηση όλων των στοιχείων. Διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να είμαστε συνεκτικοί για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την αγορά. Γι' αυτό το λόγο καταθέτηκαν και τόσες τροπολογίες, αλλά μας έδωσε κάποιες οδηγίες η συγγετρία. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχει και πάλι λέω ιδιαίτερη ακρίβεια σαφής ορισμός, επαναλαμβάνω, των πρακτικών στις οποίες, ε, οι οποίες είναι αποδεκτές από τις αγορές. Δεδομένου ότι υπάρχουν πάρα πολλέ μεγάλες και δομικές αλλαγές. Από όσον καταλαβαίνω θα πρέπει η νομοθεσία αυτή να είναι ε, συμπεριληπτική και των ε, νομοθεσίες και των αγορών και των διαφορετικών τύπων συναλλαγών. Γι' αυτό το λόγο συμφωνώ με την ε, να συμπεριλάβουμε εδώ και τις προσπάθειες χειραγώγησης των αγορών, όπως ανέφερε η συγγήτρια. Διότι νομίζω ότι το θέμα αυτής της απόπειρας χειραγώγησης ε, δεν θα πρέπει να συμπεριληφθεί. Δεν θα πρέπει να βλέπουμε μόνο χειραγώγηση και τις απόπειρες που γίνονται. Επίσης, κάτι άλλο το οποίο μας απασχολεί είναι αυτό το οποίο πραγματικά προστατεύονται κάποιες τροπολογίες για τον πολλαπλασιασμό των κυρώσεων. Έχουμε στον τομέα αυτό πάρα πολλούς ε, κανόνες, ε, αλλά υπάρχουν παντού κενά. Θα πρέπει αυτά να διορθώσουμε και θα πρέπει να μην πολλαπλασιάζουμε τις κυρώσεις, γιατί ε, κυρίως όσον αφορά τις ΜΜΕ, όπως είπε και η, η συγγήτρια η διαφορά μεταξύ μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων ε, είναι ότι είναι μικρές. Άρα θα πρέπει να το λάβουμε αυτό στο, το στοιχείο υπόψη. Ε, αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιες από αυτές δεν διαθέτουν τέτοιου είδους πληροφορίες. Θα πρέπει να είμαστε λοιπόν πολύ προσεκτικοί στη διατύπωση αυτή. Τώρα, επαναλαμβάνω, εμείς Έχουμε πάρα πολλά νομοθετήματα όσον αφορά τα θέματα των ε, κυρώσεων, αλλά έχουν πάρα πολλά κενά επαναλαμβάνω. Αυτό θα πρέπει να διορθωθεί και πάλι επαναλαμβάνω. Και να μην προβλέψουμε πάρα πολλές εξαιρέσεις και πολλαπλασιών των εξαιρέσεων. Τώρα, οι OTCs, αυτού του είδους οι συναλλαγές οι εξωχρηματιστηριακές θα πρέπει να είναι συναλλαγές τις οποίες θα υπακούν σε όλα τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί μέχρι τώρα. Και θα πρέπει να προσπαθήσουμε τα κενά, τα παραθυράκια στην ε, νομοθεσία να τα διορθώσουμε, όχι να δημιουργήσουμε ακόμη περισσότερο, διότι νομίζω ότι στον τομέα αυτό της αγοράς υπάρχουν ήδη αρκετά προβλήματα. Επίσης πιστεύω ότι θα πρέπει να εντοπίσουμε πιο περιοριστικούς τρόπους με τους ε, οποίους ε, δεν θα επιτρέψουμε να διεξάγονται και να αναλαμβάνονται δραστηριότητες που είναι μόνο επιζήμιες για τις αγορές. Επίση, θα πρέπει να επιστήσει ιδιαίτερα την προσοχή μας στο θέμα της κοινωνικής διάστασης κάποιων αγορών που πρέπει να προστατεύσουμε. Τώρα, οι ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση και να μπορούν να μοιράζονται μεταξύ του όλες τις διαθέσιμε πληροφορίε. Πάρα πολλέ φορές ε, επαναλαμβάνω, έχουμε υιοθετήσει νομοθεσία που έχει καλή πρόθεση αλλά σιγά σιγά είναι, ε, αποβαίνει περιοριστική για τις ρυθμιστικές αρχές και τους ζητούμε να κάνουν κάτι το αδύνατο. Πώς θα το κάνουν αν δεν έχουν πρόσβαση στις κατάλληλες ε, ε, πληροφορίες. Αυτό είναι κάτι το οποίο οδηγεί στις καταχρήσεις εκ μέρους των αυτών που διαθέτουν πληροφορίες στις αγορές. Αυτό είναι σημαντικό. Πιστεύω και πάλι ότι θα πρέπει να δούμε την ε, νομοθεσία. Θα πρέπει καλή να προβλέψουμε οι ρυθμιστικές αρχές να έχουν ε, ε, καλύτερα περισσότερες προφορίες παρά λιγότερες για να μπορούν να ενεργούν με τον κατάλληλο τρόπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ δεν θα μιλήσω. Και για να ολοκληρώσουμε, δίνουμε και πάλι το λόγο στην Αρλίν. Πρέπει την συζήτηση να την ε, ολοκληρώσουμε τώρα γιατί μετά έχουμε και το θέμα του προϋπολογισμού του 2013. Πολύ σύντομα. Τι θέλω να πω, ότι πρέπει να συζητήσω περαιτέρω με τους Κιώδης, να βρούμε κάποιες εναλλακτικέ λύσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις πάρα πολύ θετικές πληροφορίες που ε, έδωσαν ε, και θα ήθελα να πω ότι ο κύριος Κονφά κατέθεσε την ε, τροπολογία εκ μέρους της ομάδας σας για αυτά τα θέματα με τα οποία εσείς αναφέρετε. Ακούστε, είναι νέος τρόπος συνεργασίας αυτό. Τέλος πάντων. Τι θέλω να πω τώρα. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες τώρα. Διότι ακούστηκαν οι παρατηρήσεις, οι ενδιασμοί κάποιων. Δεν έχουμε χρόνο και εγώ πρέπει να φύγω και να δω για την οδηγία της διαφάνειας κάποιους εκπροσώπους του Σουδάν και από την Ουγκάντα και δεν θέλω να με περιμένουν. Δεν νομίζω ότι μπορούμε ούτως ή άλλως τώρα να συζητήσουμε πλήρως το θέμα αυτό των ποινικών κυρώσεων, διότι μόνο πολύ πρόσφατα μπορέσαμε να καταλήξουμε με τη Λίμπε Συμφωνία, άρα θα πρέπει να παρατείνουμε την προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών για αυτά τα θέματα. Εκτός από το θέμα λοιπόν των ορισμών, όλα αυτά τα θέματα θα τα εξετάσουμε, τα υπόλοιπα θέματα θα τα εξετάσουμε μαζί με τη ΛΥΜΠΕ. Και δεν μπορώ σε πέντε λεπτά να αναφερθώ σε ένα θέμα που χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Απλώς θα ήθελα σαν να πω ότι Εάν ολοκληρώνεται εδώ η συζήτησή μας, με τους συναδέλφους, τους κοιόδης συζητητής θα συζητήσω για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμβιβαστικές λύσεις. Θα συζητήσουμε και θα δούμε και με τον κύριο Φέρμπερ τα θέματα τα κοινά με το ΜΙΦΙΤ και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε πλειοψηφικά σε συμφωνία. Βλέπω ότι η συγγήτρια της ΛΥΜΠΕ ε, θέλει το λόγο. Αποφασίσαμε ε, να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Μόνο ένα λεπτό αν θέλετε να πείτε κάτι σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το ερώτημά μου είναι πολύ πρακτικής φύσης. Και εγώ θέλω να γίνει και στην Επιτροπή μας και εδώ η συζήτηση. Το ερώτημα μου είναι αν η προθεσμία ε, θα παραταθεί. Μπορείτε να μας δώσετε κάποια νέα. Διότι όπως ξέρετε ήταν πάρα πολύ σφιχτά τα πράγματα όσον αφορά τις προθεσμίες στην ΛΥΜΠΕ. Θα θέλαμε περισσότερο χρόνο αν είναι δυνατόν. Τώρα, τώρα έφτανα στο χρονοδιόγραμμα. Από όσον βλέπω, το ΜΙΦΙΤ θα συζητηθεί πρόταση με τον κανονισμό. Άρα θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ψηφίσουμε τον Ιούλιο στην συνεδρίαση και στην Ολομέλεια το Σεπτέμβριο και εγώ θα δω πώς έχουν και τον άλλον τα χρονοδιαγράμματα και οι προθεσμίες ώστε να μπορέσουμε να αλλάξουμε και να παρατείνουμε την προθεσμία και θα πρέπει να δούμε και σε συνεργασία με τις άλλες επιτροπές και τους συναδέλφους τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Και ήθελα να σας ευχαριστήσω για την κατανόησή σας ιδιαίτερα σε αυτούς, αναφέρομαι σε αυτούς που περιμένουν και το, να λάβουν το λόγο για το θέμα 10, για τον προπολογισμό δίδω Το λόγο στον εισηγητή και όπως μας είπαν και οι διερμηνείς μπορούμε να μείνουμε και 10 λεπτά παραπάνω αν χρειάζεται. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αρχίζοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τη γραμμαρία και το προσωπικό που με βοήθησε να κάνω αυτή την ε, σχέση. Αυτό το, με το σχέδιο γνωμοδότησης. Εμείς ξέρετε ότι όσον αφορά την διαδικασία, μετά την πρόταση της Επιτροπής, ε, καταθέτουμε τροπολογίες, ε, παρουσιάζεται το πρώτο ε, θέμα αυτό στον Ιούλιο. Μέχρι τις 24 Ιουλίου έχουμε τρο, προθεσμία εμείς για να καταθέσουμε τροπολογίες. Όπως ξέρετε, για να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη στις αγορές και να υπάρχουν ισορροσκημένοι προϋπολογισμοί θα πρέπει να προχωρήσουμε φέτο. Καταλαβαίνετε ότι τα προβλήματα στις χρηματοπιστωτικές αγορές, η αύξηση του δανεισμού, ε, η αύξηση ε, θα πρέπει κάτι να κάνουμε και ενδεχομένως να αυξήσουμε και τη φορολογία. Αυτό είναι κάτι το οποίο απασχολεί όλους τους ε, πολίτες μας. Ξέρουμε ότι πριν από δύο χρόνια το επιτόκιο δεν ήταν 4% τώρα ξεπερνάει το Το Ξέρω να επιδείξουμε αλληλεγγύη, αλλά η αλληλεγγύη είναι απαραίτητη και άρα χρειάζεται να γίνει η διαπραγμάτευση του προπολογισμού. Θα πρέπει λοιπόν το Κοινοβούλιο να επιδείξει και αλληλεγγύη σχέση με του φορολογούμενου. Και θα πρέπει το Συμβούλιο να το εκλάβουμε ω ε, συνομιλητή και όχι ω ανταγωνιστή. Θα πρέπει να μπορέσουμε να ιεραρχήσουμε και εμείς την ε, ε, δαπάνες και να είμαστε θετικοί μόνο εκεί, το οποίο, εκεί όπου μπορούμε να προβλέψουμε ε, ανάπτυξη. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε έναν προεπισμό τη τάξη του 1% του δικού μα. Σωστά λέγεται ότι οι περικοπές του κοινοτικού προπολογισμού δεν θα επιλύσουν την κρίση αλλά και δεν θα βοηθήσει υπερβολικά τα κρατημέλη. Σωστό. Αλλά μία αύξηση κατά 7% στο προπολογισμό επίση δεν θα ε, αλλάξει και εκβαθέν την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η πρόταση που κάνουμε είναι να... Ε, ε, αυτή η πρόταση είναι να κάνει να φαίνεται εντελώς ε, γελία η Επιτροπή στη σημερινή ε, εποχή. Αυτό το οποίο θέλω εγώ να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε ότι κάνουμε στις χώρες μας που ζητούμε λιτότητα και δημοσιονομική πειθαρχία να το ζητήσουμε και από την Επιτροπή. Βεβαίως είναι περιορισμένες οι αρμοδιότητες μας, αλλά θα πρέπει να μπορέσουμε να κάνουμε περικοπές που θα μας επιτρέπουν να κάνουμε εκεί που χρειάζονται κάποιες αυξήσεις. Θα πρέπει στην, εμείς, την Επιτροπή Προεπιλογισμών και το Συμβούλιο να παρουσιάσουμε ορθολογισμένες προτάσεις και για την άποψή μας θα πρέπει να ε, ζητήσουμε πάγωμα κάποιων τιμών. Είμαι ο Σκιώδης συγητής της ομάδας μου για το Omnibus 2 και για το CIA 3 και έχω καταθέσει πολλές τροτολογίες για την CIA 4. Εδώ ζητούμε να ε, δοθούν στην ίσες νέες αρμοδιότητες και να μπορέσουμε σε θέματα αυτά να δώσουμε προτεραιότητα σχέση με τις υπόλοιπες γραμμές. Κάθε φορά που ίσεις ή άλλοι οργανισμοί ε, ε, αναλαμβάνουν νέα καθήκοντα, θα πρέπει να τα συνοδεύουμε με τα κατάλληλα κονδύλια. Αν θέλουμε να είμαστε υπό, υπεύθυνοι θα πρέπει τις προτάσεις που κάνουν τις συνοδεύουμε και με τα καλά τα κονδύλια. Η θα πρέπει να είναι αντικειμενική δεδομένου ότι μόνον έτσι δεν είναι αποτελεσματική. Πρέπει λοιπόν να δούμε ποια είναι τα διαφορετικά χρηματοδοτικά μοντέλα τα οποία θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε και το άχθος από τους προλογούμενους. Πριν όμως θα πρέπει να δούμε πώς έχει το χρηματοδοτικό πρότυπο το οποίο ακολουθούμε. Για να μπορέσουμε λοιπόν να καταβάλουμε τα κατάλληλα ε, ε, κονδύλια ε, για να μπορέσουν ε, να φέρουν σε πέρα στα επιπρόσθετα καθήκοντά τους οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, θα πρέπει να δούμε την ε, γραμμή κρίνης του προϋπολογισμού που ασχολείται με αυτά τα θέματα. Εδώ προτείνει για του χρόνου 5 εκατομμύρια ευρώ η Επιτροπή παρά το γεγονός ότι πέρσι υποχρεώσεις πληρωμών έφτασαν μόνο στο 4 εκατομμύρια. Και παρά το γεγονό ότι πέρσι στην ίδια γραμμή του προπολογισμού χρησιμοποιήθηκαν 79 εκατομμύρια, προβλέπει 100 η Επιτροπή. Επίση, σε θέματα ε, Ένωση, νομίζω ότι μπορούμε επίση να κάνουμε αποταμίευση, δεδομένου ότι υπάρχουν. Με συγχωρείτε, ε, ε, στα φορολογικά θέματα νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε οικονομίε, δεδομένου ότι αντιτίθεται πολλά κράτη-μέλη εδώ και πάλι θα πρέπει να γίνει ράση προτεραιοτήτων. Και θα ήθελα να υπάρχουν συμπληρωματικά κονδύλια για τις προτεραιότητες, εάν ε, πολλά μέλη συνοδεύουν αυτές οι προβλεπόμενες αυξήσεις με κάποιες ε, περικοπές. Εμείς στην ΕΚΟΝ θέλουμε ε, να πούμε ότι όντως υπάρχουν ε, περιθώρια αύξησης κάποιων κονδυλίων και εγώ θα ήθελα να συνεργαστώ με συναδέλφους άλλων ομάδων για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια συνενετική λύση. Ευχαριστώ. Ο Ζαμπόλ που ήρθε προηγουμένως έφυγε αλλά εκ μέρους των σοσιαλιστών δίνω στον συνάδελφο το λόγο. <clears throat> Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για αυτό το σχέδιο της έκθεσης. Νομίζω ότι πραγματικά όταν μιλάτε για τις ε, προτεραιότητες έχετε χτυπήσει φλέβα. Για την πλευρά της ΕΚΟΝ είναι σημαντικό να ε, διασφαλίσουμε ε, τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών ε, εποπτικών αρχών. Απλώς βρισκόμαστε μπροστά σε ένα σταυροδρόμι. Οι αρχές μιλάνε για αύξηση του προϋπολογισμού έως και 40% για να κάνουν αποδοτικά και αποτελεσματικά τη δουλειά τους. Νομίζω ότι αυτό είναι ε, πολύ σοβαρό ποσό εκτίμηση, ε, αλλά ε, τα ε, καθήκοντα που θα τους ε, αναθέσουμε είναι πολύ πολύ πλοκά. Είναι δύσκολο λοιπόν κανείς να διατηρήσει την ποιότητα χωρίς να διαθέτει επιπρόσθετους πόρους. Πέρα, παρά από αυτό όμως η Κομισιόν προτείνει ένα μίνιμουμ αύξησης για το EBA και επίσης μια σειρά μειώσεων για την ΕΑΚΑ και το IOPA. Ε, είναι δύσκολο να παρακολουθήσουμε τη λογική ε, εξαγωγή συμπερασμάτων ε, στον τρόπο που σκέφτεται η Κομισιόν. Νομίζω ότι η χρηματοδότηση παίζει ρόλο προς τις ικανότητες των εποπτικών αρχών. θέλουμε πιο ισχυρές αγορές, γι' αυτό χρειαζόμαστε και ισχυρότερη, όχι πιο ασθενή ε, εποπτεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο εισηγητής μιλάει για ένα άνοιγμα σε ένα χρηματοδοτικό ε, μοντέλο όπου οι παίκτες οικονομικοί θα συμβάλλουν και αυτή ε, στιγματοδότηση των αρχών. Νομίζω ότι σε κάποια κράτη-μέλη αυτό λειτουργεί καλά. Θα μπορούσε να λειτουργήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο εισηγητής έχει απόλυτο δίκαιο στις ε, βασικές του προτεραιότητες. Όμως, όταν φτάνουμε σε συγκεκριμένα ε, σημεία, έχω κάποια ερωτηματικά. Ήμασταν ε, πολύ περιοριστική ε, ως προς τη δημοσιονομική μας δουλειά, αλλά αν είμαστε κατηγορηματικοί ως προς το πάγωμα του προϋπολογισμού. Μάλλον πάμε λίγο μακριά. Μιλάμε για ε, μια προσπάθεια να ταιριάζουν οι δραστηριότητες με τους πόρους. δεν πρέπει εξ αρχής να θέτουμε λοιπόν πλαφόν γιατί αυτό θα μπορεί να βλάψει σημαντικά ε, τις δραστηριότητες. Υπάρχουν κάποια σημαντικά στοιχεία που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας. Όταν εσωτερικά η Κομισιόν ε, αντιμετωπίζει το θέμα της ε, οικονομικής διακυβέρνησης, στην Κεντρική Διεύθυνση Εξφένη υπάρχουν αρκετοί πόροι για να μπορέσουν να εκτελεστούν τα απαραίτητα καθήκοντα υποπτίας του προπολογισμού. Τα δύο πακέτα θα εφαρμοστούν μέχρι το φθινόπωρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει όλο και περισσότερους ε, χειριστές που θα, που θα ε, λειτουργούν εντός του συστήματος. Ε, ε πώς ε, θα διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν κατάλληλα κονδύλια για αυτούς. το θέμα λοιπόν των διοικητικών δαπανών είναι ένα ζήτημα που πρέπει να θέσουμε. Ένα άλλο ζήτημα που ήθελα να ανοίξω είναι οι στατιστικές. Περνάμε από το ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα στο άλλο. Πρέπει να βρούμε το κατάλληλο επίπεδο κονδυλίων. Στην Ευρώπη οι στατιστικές έχουν όλο ένα και μεγαλύτερη σημασία για τη διατήρηση της βιωσιμότητας είναι σημαντικό ε, όσον αφορά στην αλληλεγγύη μεταξύ των εφορολογουμένων. Είναι σημαντικό λοιπόν οι αρχές να μπορούν επαρκώς να εκτελούν τα καθήκοντά τους. Έτσι λοιπόν ε, προσβλέπω σε μια επικοδομητική συζήτηση και θέλω πραγματικά να δω ε, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα τις επόμενες ημέρες. Ευχαριστώ. Καρλ Χέγκλαντ είναι ο σκιώδης του Άλντε που έφυγε για να γίνει ε, υπουργό, άρα εγώ θα ε, έλθω ως αντικαταστάτρια. Χαιρετίζω τα όσα κάνατε, ειδικότερα την ιδέα ε, της ε, θέσπισης προτεραιοτήτων. Είναι κάτι το οποίο όλοι θα προσυπογράψουμε. Είναι σημαντικό που θα μπορέσουμε να βρούμε σημεία στα οποία μπορεί να γίνει εξοικονόμηση χρηματοδότησης. EBA ε, παίρνει περισσότερα χρήματα γιατί ε, θα έχει περισσότερη δουλειά στο CRD. Η ΕΚΑ είναι καλύτερα από τους άλλους γιατί ήδη παίρνει χρήματα από τη βιομηχανία γιατί χρεώνει ε, ο ρόλος της για, τις, ε, για τα γραφεία αξιολόγησης, τους οίκους αξιολόγησης. Οι αιώπα, ας πούμε, έχουν πολύ σημαντικές δυσκολίες και λόγω κάποιων ε, κακών ε, υπολογισμών, δηλαδή δεν υπολογίζουν σωστά ε, το προσωπικό τους. Τέλος πάντων, υπάρχουν πολλά τέτοια σημεία. Φαίνεται ότι όλα αυτά επιβαρύνουν την ΑΙΟΠΑ. Όμως, ε, στον προπολογισμό μισθοδοσία, για παράδειγμα. 7.890 για το 2013, το οποίο είναι σταθερό σε σχέση με το 2012 και δεν ε, έχει νόημα αυτό γιατί είχατε πει ότι υπάρχουν 21 εκατομμύρια για τη μακροοικονομική αρρωγή. Ίσως θα μπορούσαμε να τα δώσουμε στην ΑΙΟΠΑ και αυτό να μην επιβαρύνει πολύ τη μακροοικονομική οικονομική υποστήριξη. Επίσης η DG ECFIN, η Γενική Διεύθυνση ΕΚΦΙΝ έχει μεγάλη πίεση με τη δουλειά που έχει να κάνει. Ίσως λοιπόν θα πρέπει να δούμε ε, πιο γενικό, την πιο γενική γραμμή του προϋπολογισμού σχετικά με τους ε, φορείς σε επίπεδο Επιτροπής Προϋπολογισμού, ε, έτσι ώστε να προσθέσουμε κάποια άλλα στοιχεία, να συμπεριλάβουμε αυτό το θέμα, ε, καθώς ε, αυτοί θα συνεχίσουν να μεγαλώνουν, θα τους δίνουμε όλο και περισσότερα καθήκοντα, από τη στιγμή που δίνουν και στη Γενική Διεύθυνση ε, ΕΚΦΙΝ πολλές ε, αρμοδιότητες και ευθύνε, νομίζω ότι θα επιβαρυνθεί το, το πρόγραμμά τους. Λοιπόν, ε, αυτά είχα να πω. Επόμενος είναι ο Σβέν. Υπάρχει μια ολόκληρη σειρά από θέματα. Βεβαίως, μέχρι στιγμής οι συζητήσει για το προπολογισμό στην Οικονομική Επιτροπή βασίστηκαν στα θέματα τα οποία καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε τώρα η συζήτηση που διεξάγεται είναι πιο φιλοσοφική και αφορά τον ε, προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι καλύτερα να, μην αφαιρθούμε σε μεμονωμένα κονδύλια που δεν παίζουν τόσο σημαντικό ρόλο σε σχέση με όλο τον προϋπολογισμό. Το πραγματικό θέμα για το μέγεθος του προπολογισμού ξέρουμε ότι είναι τα διαδροτικά ταμεία, η γεωργία και βεβαίως εκεί μπορεί να υπάρχει μία αιτιολογημένη άποψη από την άποψη Οικονομικής Επιτροπής. Ας συζητήσουμε όμως αυτά τα θέματα, γιατί υπάρχουν και οικονομικές προεκτάσεις. Θα πρέπει όμως να συζητήσουμε κατά πόσον το κοινό νόμισμα χρειάζεται αυτόματους σταθεροποιητές, καθώς και τι ρόλο θα μπορούσε να έχει ένα ένας ενδιαμβωμένος προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταλαβαίνω ότι ο προπολογισμό δεν είναι τόσο αποτελεσματικό στην εξυπηρέτηση αυτού του ρόλου. Συνεπώς χρειαζόμαστε τη διεξαγωγή μιας συζήτησης σε μακροοικονομικό επίπεδο. Και πραγματικά ελπίζω ότι όταν καταλήξουμε σε μια κοινή γνωμοδότηση θα επανέλθουμε και πάλι στα σημαντικά θέματα που καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε και θα προσπαθήσουμε να αποφύγουμε μια εκτενή ιδεολογική συζήτηση και μετά θα περάσουμε στην ε, ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Βεβαίω η ίδια συζήτηση θα πρέπει να διεξαχθεί και ε, πάλι, ε, εγώ πραγματικά είμαι πνιγμένο στο, στο νομοθετικό μου έργο, αλλά σε κάθε περίπτωση ελπίζω να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εκδοχή της έκθεσης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα θέματα, είναι καλό το ότι το ότι χρειαζόμαστε περισσότερα ε, χρήματα Θα πρέπει να πω ότι με απογοήτευσε το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν ανταποκρίθηκε στα αιτήματα σας. Ήταν αρκετά λογική, υιοθέτησαν μια αρκετά λογική στάση σε ό,τι αφορά τις πράξεις κατεξουσιοδότησης. Ε, και εξουσιοδότηση. Πολύ λογική. Επιτροπή απαντάει σε αυτό με μία μείωση στον προπολογισμό ΕΣΜΑ και ΙΟΠΑ σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο και δεν ε, λαμβάνει υπόψη τα αιτήματά τους. Ε, αυτή είναι η... Την αντίθεση δεν την περίμενα από πλευρά τη Επιτροπή. Δεύτερον, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα στο θέμα χρηματοδότησης. Από τη στιγμή που δεν έχουν μία, έναν εξάρτητο κονδύλιο, η Επιτροπή έχει πάντοτε το κίνητρο να μειώσει, να περιορίσει την ε, ε, το προπολογισμό του ΕΣΑΣ. Νομίζω λοιπόν ότι θα υπάρξει μια ανεξάρτητη γραμμή του προπολογισμού. Ύστερα το θέμα των ε, εναλλακτικών πηγών χρηματοδότηση. Θα πρέπει να πω ότι ξέρουμε ότι η ΕΣΜΑ ε, έχει λιγότερα προβλήματα γιατί μπορούν να βρουν κονδύλια για την εποπτεία των οργανισμών ψελιπτικής ικανότητας. Βεβαίω Υπάρχει κάποια βάση αυτό. Θα πρέπει όμως να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να μην κάνουμε λάθη. Ε, επειδή η βιομηχανία θα πρέπει να ε, ε, επιβάλλει κάποιο τίμημα, θεωρεί ότι έχει και ένα ρόλο. Θα πρέπει να υπάρχει η αρχή του διαχωρισμού μεταξύ του ρόλου του εποπτεύοντος κράτους και της βιομηχανίας. Ξέρω από την Γερμανία τον ατυχή ρόλο της βιομηχανίας, στους εποπτικούς φορείς. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι είμαστε σαφώς υπέρ της πρότασης του Κοινοβουλίου για το φετινό προπολογισμό για να υπάρξει αύξηση των δαπανών σε το τομέα διεθνούς συνεργασίας. Είμαστε κατά του ότι δεν συμπεριλήφθη αυτό στον προπολογισμό. Αυτό ήταν ένα επίτευγμα του Κοινοβουλίου και θα πρέπει να ε, συνεχίσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεν υπάρχει αιτιολόγηση για τον περιορισμό των δαπανών στην ε, επιβολή φόρων. Ορισμένες χώρες διαφωνούν και αυτή είναι η βασική φιλοσοφία που θα αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Ένωση με ή χωρίς μερικά από τα μέλη. Και αυτό βεβαίως υποστηρίζει μια μεγαλύτερη ολοκλήρωση και δεν μπορεί να αποτελέσει αιτιολόγηση για διακοπή της συνεργασίας σε ένα τόσο σημαντικό τομέα. Ευχαριστώ. Θα δώσω τον υπόλοιπο χρόνο που μας έχουν δώσει διερμηνείς στον ΣΑΜ και μετά θα συνεχίσουμε μεταξύ μας αγγλικά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα πω το εξή σε δύο λεπτά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαιρετικό σχέδιο γνωμοδότηση. Η ευρωπαϊκή οικονομική κρίση συνεχίζεται και για να είμαστε αξιόπιστοι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι σε επίπεδο και κρατών μελών και θεσμικών οργάνων θα πρέπει και φορολογωμένων οι πάντες να λάβουν υπόψη ότι δεν ενεργούμε με λόγια, αλλά και με έργα και με αριθμούς. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε σε σαφήνεια με όλους ότι δεν ζούμε απομονωμένοι εμείς στη, στο πλανήτη μας και ξέρουμε ποια είναι τα καθημερινά προμήθεια. Εάν θέλουμε περισσότερα χρήματα, θα δυσφημιστούμε. και δεν θα πάρουμε και χρήματα. Είμαι λοιπόν υπέρ τη γραμμή που υιοθέτησε ο εισηγητή όσον αφορά το πάγωμα του προπολογισμού και θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στην ανάπτυξη και να εξασφαλίσουμε το ότι όταν θα αυξήσουμε κάπου, κάπου θα πρέπει να περικόψουμε στον προπολογισμό. Ευχαριστώ, ευχαριστώ τους διερμηνείς και δίδω το λόγο στον Ashley.